Now. Please take your seats. Please take your seats. Καθίστε παρακαλώ. Dear colleagues, we are about to have an electronic vote. Συνάδελφοι, θα ψηφίσουμε το σημείο 12 ηλεκτρονικά για το ε, κατάταξη των τρίτων χωρών, των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να έχουν στην κατοχή τους θεωρήσεις όταν ε, περνούν τα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών και των οποίων οι, ε, και των οποίων οι υπήκοοι εξαιρούνται από αυτή την απέτηση. Λοιπόν, πάμε στην ψηφοφορία. Amendment number one. Τροπολογία 1. The vote is open. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Excuse me, it didn't work. Τι έγινε, δεν δουλεύουνε τα συστήματα. How many of you? Για πόσους δεν δουλεύουν, πόσοι δεν ψηφίσατε ηλεκτρονικά. Θα την θα ξαναψηφίσουμε. Αλλάξατε θέσεις όσοι δεν ψηφίσατε πριν. We're going to reopen. Amendment 1, Recital 9 Τροπολογία 1. Εκτελογική σκέψη 9α. Now the vote is closed. ψηφοφορίας. Δεν, λειτουργεί. Μπορείτε να αλλάξετε θέση, να κάτσετε πιο δίπλα. Ε? Yes. Two votes in favor, 49 against, so it's rejected. Δύο υπέρ, 49 κατά. Άρα Απορρίπτεται. Συνολική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. «49 υπέρ, 2 κατά». Εγκρίνεται η έκθεση. Η κυρία Φαγιόν θέλει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις συγητές και τους ε, συναδέλφους για την υποστήριξή τους και σύντομα να πω ότι θα στείλουμε ένα πολύ θετικό και πολύ έντονο μήνυμα στις χώρε ε, στις ε, χώρες ότι, στην Βοσνία Ζεγοβίνη και στην Σερβία ότι μπορούμε να άρουμε την υποχρέωση για τις θεωρήσεις. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο και άλλες χώρες ώστε να μπορέσουμε σύντομα να ολοκληρώσουμε την όλη διαδικασία. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ κυρία Φαγιόν και συγχαρητήρια. Και την συγγήτρια, την κυρία Κοράτσα Βίλτ. Πάμε σε δεύτερη ψηφοφορία. Πριν όμως προχωρήσουμε για την ενιαία διαδικασία υποβολής ε, αίτηση για τη χορήγηση άδεια διαμονή και εργασία. Η κυρία Μπατία θέλει το λόγο. <laughs> Euh, Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δύο προφορικέ τροπολογίε. πιστεύω πω το έχετε. Στο άρθρο 3 δεν θα το αναφέρω συγκεκριμένα, αλλά να σας πω ότι είμαι ευτυχής που η έκθεση αυτή θα είναι ενώπιον της Επιτροπής σήμερα, γιατί είναι η τρίτη φορά που παρουσιάζει η Κομισιόν αυτό το αίτηση για ενιαία άδεια ε, και να ευχαριστήσω τους και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν, να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία και αυτά. Νομίζω πως φτάσαμε σε διάφορες συμβιβαστικές τροπολογίες μετά από πολλούς μήνες πραγματεύσαν και ας ψηφίσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Παδία. Ε, πάμε στην ψηφοφορία. Τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. No. Not working. Now, now, now the vote is open. The vote is... Τώρα άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας. 45 υπέρ, 4 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Now the vote is closed. Πέρας. Είχαμε και 47 υπέρ, μία ψήφος κατά. Άρα εγκρίνεται. Με ανάταση της χειρός θέλετε να ψηφίσουμε. Εντάξει. Άρθρο, συγγνώμη, τροπολογία 6. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 17. Συγγνώμη. 18. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 7. Τροπολογία. όχι 7. Συγγνώμη. Προφορική τροπολογία του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Τροπολογία 82. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Τροπολογία 86. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Απορρίπτεται. 87. Όχι. Συμβιβαστική πρόταση 4. Υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Oral amendment. Amendment 32. 32. Υπέρ. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. 25. Υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Όχι, εγκρίνεται. Να το ελέγξουμε καλύτερα. Για να το ελέγξουμε. Τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 33 υπέρ και 17 κατά. Εγκρίνεται. 26. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται, ε. Να το ελέγξουμε. Για να το ελέγξουμε. Τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας. 32 υπέρ, 19 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 27. 27. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται. Σας παρακαλώ όμως λίγο να κρατάτε τα χέρια σας ε, ψηλά γιατί καμιά φορά δεν ε, είναι σαφές. Τροπολογία 93. Υπέρ. Against. Κατά. Amendment 90. Υπέρ. Τροπολογία 90. Τροπολογία 90. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για το άρθρο 3. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 5. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 40. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 41. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 41. Να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Now what is closed. Πέρας ψηφοφορίας. So it's 25... 22 υπέρ, 25 κατά. Απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά. Νομίζω απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέρας. 23 υπέρ, 26 κατά. Απορρίπτεται. Ε, τροπολογία 44. Υπέρ. Όχι. Λάθος. Λάθος, λάθος. Βιάζομαι. Τροπολογία 99 υπέρ κατά απορρίπτωτο Τροπολογία 44 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 6 υπέρ κατά εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 7 υπέρ κατά Να το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Board is closed. Πέρας 24 υπέρ, 27 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Λάθος. Ε, τροπολογία 48. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ. Βιάζεται ο πρόεδρος. Κατά. Νομίζω εγκρίνεται. Δεν ήταν σαφέ τι έγινε με το συμβαστική 8. Πάμε πάλι στη συμβαστική 8 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Α, να το, για να το ελέγξουμε. Για τη συμβαστική 8 ψηφίζουμε. 26 favor, 20... 26 υπέρ, 24 κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ. Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. κατά εγκρίνεται 104 υπέρ κατά να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά 104 Now, I voted. Uh, excuse me. No, I got I got my my my voting list. 104. 20 υπέρ, 31 ψήφι κατά. Απορρίπτεται. 105 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. Απορρίπτεται. Συμβαστική εννέα. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία. Okay. Second part. Yes. The second part of a Δεύτερο τμήμα της 106 ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 106. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 52. Υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε. Την 52 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μα έχω τον κατάλογο μπροστά μου. Όχι, μετά θα τα διορθώσω αν τα λέω λάθος. Well, even up my vote Εντάξει, ακόμη και αν σε όλες ψήφισα αρνητικά, το αποτέλεσμα είναι 29 προς 22. Κάτι γίνεται, μάλλον έχω λάθος ε, λίστα ψηφοφορίας, τι να σας πω. Κάτι συμβαίνει πολύ άσχημα πάντως. Okay, okay, okay, okay. Okay. Now,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 Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 53. Όχι. There are three positions. Yes, no, and abstention. That's the position of the rapporteur. Okay, okay. They should have your, your voting. Now, the vote is closed. Πέρα ψηφοφορίας. 33 favor 31 ε, ψήφοι υπέρ και 18 κατά εγκρίνεται. 109. Όχι. Καταπίπτει. Εκατόν δέκα. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 111. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 55. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά εγκρίνεται νομίζω 112 ε, υπέρ κατά απορρίπτεται 114 υπέρ Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. 57. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 58. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. 59 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. 59 ηλεκτρονικά. No. Closed. 31 ψήφοι υπέρ, 20 ψήφοι κατά ήταν το αποτέλεσμα. Εγκρίνεται η τροπολογία. 116 υπέρ κατά απορρίπτεται 118 υπέρ 117 υπέρ συγγνώμη 117 υπέρ κατά Απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται νομίζω. 119. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 60. Board is closed. Πέρας. 34 ψήφια υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 120 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η 121 αποσύρεται. 64 υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίζουμε την 64. Vote is Πέρας ψηφοφορίας. 28 υπέρ, 20 κατά. Εγκρίνεται. Πάμε σε τελικές σκέψεις. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 65. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 66 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Για να το ελέγξουμε. Τροπολογία 2. Vote 30. Πέρας. 30 προς 21. Εγκρίνεται. Συμβαστική πρόταση 10. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Τροπολογία 3. Τροπολογία 3. Τροπολογία 3. Υπέρ. Η τροπολογία 3 παραμένει. Τροπολογία 3, αν δεν κάνω λάθος, παραμένει. Ψηφίζουμε την 3 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την 3. Board is closed. Πέρασε ο 24 προς 25. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ ε, δεν είναι σημαντικό, αλλά μήπως μπορείτε να φωνάζετε και τις αποχές, γιατί έχουμε και αρκετές αποχές κάθε φορά. Ε, ναι, εντάξει, έχετε δίκιο, αλλά απλώς για να πάμε λίγο γρήγορα. Ε, εντάξει, αν θέλετε φυσικά θα ζητώ και τις αποχές. Συμβιβαστική 13 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ορίστε. Εντάξει κύριε Ταβάρης. Ζητώ συγγνώμη, ταπεινά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10. Υπέρ κατά αποχές να το ελέγξουμε ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη 10 Vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας 33 προς 15 εγκρίνεται Τροπολογία 72 υπέρ κατά Απορρίπτεται. Συγγνώμη, αποχές, αποχές. Τώρα απορρίπτεται. 74. Όχι, 74. Καταπίπτει. 25 εγκρίθηκε. 75. Τροπολογία 75. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 76. Υπέρ. κατά, αποχές, απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, αποχές, για να το ελέγξουμε. Ψηφίζουμε χρονικά την 11. Boris closed. 37. Πέρας. 37 προς 14. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 78 σε δύο τμήματα. Ψηφίζουμε το πρώτο τμήμα. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79, πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα, υπέρ, όχι, λάθος. Πάμε στο δεύτερο τμήμα της 79, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Αρχικό κείμενο. Ε, αιτιολογική σκέψη 19. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 8 κατά. Σας ευχαριστώ πολύ και για την υπομονή σας και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Thank you, colleagues. If you please, we move, move on. We're moving on. Congratulations again. But if you please allow us all. σας παρακαλώ, να προχωρήσουμε στο σημείο 14, στο επόμενο. Point for concerns the minimum standards. Αφορά τις ελάχιστες προδιαγραφές I beg for your attention and please to remain. Προσέξτε με παρακαλώ και Παρακαλώ να σιωπάσετε, α, να σιωπάσετε αν μείνετε στην αίθουσα, για να προχωρήσουμε στο σημείο 14. Ελάχιστες απαιτήσει για την αναγνώριση και το καθεστώς των επικών τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το παρεχόμενης προστασίας. Έχουμε εδώ να εξετάσουμε ένα έγγραφο εργασίας. Θα ακούσουμε την κυρία Λάμπερτ, η οποία... The working document. οποία θα μας παρουσιάσει το έγγραφο εργασίας για ένα πολύ σημαντικό μέσο εργαλείο του πακέτου ασύλου. Να επιστήσουμε την προσοχή σας στο ότι για να εκμεταλλευτούμε την ε, φάση αυτή που μας προσέφερε η Βελγική Προεδρία για την οποία είναι προτεραιότητα το άσυλο η κυρία Λάμπερτ παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσής της στην επόμενή μας συνεδρία στις 11 Οκτωβρίου. Ο στόχος είναι να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Βελγική Προεδρία τον Νοέμβριο αφού θα έχουμε συζητήσει το έγγραφο εργασίας και θα έχουμε ζητήσει το... και από την Βελγική Προεδρία να μοιραστεί μαζί μας ε, κάποιες πληροφορίες όσον αφορά την εξέλιξη και την πρόοδο του θέματος. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίω ε, έχουμε συζητήσεις με την Βελγική Προεδρία αμέσως μετά την απόφαση στην Επιτροπή και την πρόοδο που μπορεί, δεν μπορεί να σημειωθεί σε σχέση με άλλα μέρσα του πακέτου περί που έχουμε επιτάπητο σήμερα. Ε, το έγγραφο εργασίας που είναι το σημείο 12 στην ατζέντα ε, έχει στόχο να δώσει ένα ιστορικό στις προτάσεις που προέρχονται από την Κομισιόν. Θα θυμάστε ότι πρόκειται για μια αναδιατύπωση της οδηγίας, δεν πρόκειται για πλήρη ε, ε, μεταρρύθμιση ε, και το έγγραφο εργασία ε, υποδεικνύει που αυτό μα ε, δημιουργεί κάποια προβλήματα και από την άλλη πλευρά πιστεύω πω μπορούμε όλοι να καταλάβουμε γιατί ίσω η Κομισιόν δεν ε, έλαβε κάποια πιο ριζοσπαστικά και αποφάσει, δεν έκανε κάποια πιο ε, έλευτα βήματα από αυτά που θα θέλαμε εμεί. Λοιπόν, το έγγραφο εργασία μιλά για κάποια από αυτά τα θέματα, δηλαδή τα εκρεμή ζητήματα και όσοι διάβασαν την αξιολόγηση της μελέτης θα αναγνωρίσουν ότι κάποια από τα στοιχεία που αρχικά είχαμε παρατηρήσει δεν υπάρχουν στην αναδιατύπωση. Σύστασή μου είναι λοιπόν να δούμε τι ακριβώς ε, είναι το πιο προβληματικό. Ένα-δύο σημεία μπορούμε να τα συζητήσουμε και βεβαίως να δούμε και ποια είναι η άποψη του Συμβουλίου. Η ισχύουσα οδηγία, όπως θα θυμάστε, ασχολείται με δύο βασικά θέματα. Το ένα είναι οι όροι που πρέπει να πληρούνται ώστε ένας άνθρωπος να μπορεί να ε, λάβει το στάτους του πρόσφυγα είτε την επικουρική προστασία. Πράγμα που σημαίνει το φόβο σοβαρή βλάβη αν κάποιο έπρεπε να επιστρέψει στη χώρα παρελευσή του. Ενώ το καθεστώ του πρόσφυγα διέπεται από διεθνείς συμφωνίες και το κίνδυνο ατομικής ε, δίωξης, προσωπικής δίωξης μάλλον. Τα κράτη-μέλη προσφέρουν προστασία σε διάφορους οι οποίοι δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες, αλλά χρειάζονται πηγόντως προστασία. Όταν ε, λοιπόν αρχικά συντάχθηκε αυτή η οδηγία υπήρχε ε, χώρος ε, για τα κράτη-μέλη να το βάλουν διάφορα δικαιώματα για τους δικαιούχους επικουρικής προστασίας. Τώρα, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έχει καταστεί σαφές ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν τη διάταξη αυτή για όλες αυτές τις διατάξεις, δηλαδή δεν το χρησιμοποιούν, χρησιμοποιούν κάποιους από τους όρους. Ορισμένα κράτη-μέλη όμως τείνουν να χρησιμοποιούν την επικουρική προστασία, ενώ αυτό που θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί είναι το καθεστώς του πρόσφυγα. Και γι' αυτό και το θέμα της, ε, προκύπτει το θέμα της ευθυγράμμισης των δικαιωμάτων για τους ε, πρόσφυγες και την ανθρωπιστική προστασία ώστε δηλαδή να αποφευθούν κάποια από τα στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν σε παρενέργειες. Πράγμα που θέλουν να αποφύγουν τα κάτι μέλη. Αυτά είναι κάποια ζητήματα που έχουμε εδώ λοιπόν σε αυτό το έγγραφο εργασία. Το θέμα της αντικατάστασης στην γλώσσα της οδηγίας του καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής ε, προστασίας θέσει σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας για να θυμίσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτό και να μπούμε στην ευθυγράμμιση των δικαιωμάτων. Κάτι ακόμα που είναι ένας ακρογωνίας λήθος όσον αφορά το ξεκαθάρισμα της γλώσσας που χρησιμοποιούμε γιατί ασκήθηκε κριτική στην οδηγία γιατί βλέπουμε διαφορές μεγάλες ε, στην λήψη αποφάσεων και στην εφαρμογή αυτής της οδηγίας μέχρι τώρα είναι ένας από τους λόγους είναι γιατί η γλώσσα είναι συγκεχημένη, άλλος λόγος είναι βέβαια εντάξει η πρακτική που ακολουθείται σε κάθε χώρα αλλά η γλώσσα θα πρέπει να είναι ε, η ίδια σε όλες τις χώρες. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε να πούμε στο άρθρο 7, ότι δηλαδή οποιοδήποτε οργανισμός που ενεργεί ως προστάτης θα πρέπει να είναι σε θέση να επιβάλλει το δίκαιο. Μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο πέρα, μπορούμε να μιλήσουμε και για λογοδοσία μέσα σε αυτό το άρθρο, τόσο για τα κράτη όσο και για οποιοδήποτε άλλη άλλο φορέα που θεωρείται φορέας προστασίας. Το άρθρο 9 αφορά την ε, δίωξη και αυτό είναι ξεκάθαρο ε, στο τι προτείνει η Κομισιόν. Τώρα, εσωτερική προστασία άρθρο 8, δηλαδή ε, ο κόσμος που κινείται εντός μιας χώρας μπορεί να βρει προστασία σε κάποιο άλλο σημείο της ίδιας χώρας. και εδώ προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τα όσα λέμε, να ορίσουμε δηλαδή τι ακριβώς εννοούμε προστασία όταν ε, δηλαδή λέμε ότι μπορεί κανείς να κινείται και να εγκαθίσταται εκεί αλλά υπάρχουν και διάφορες άλλες παρατηρήσεις ε, από τον ε, UNHCR και άλλους αλλά εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να διατηρήσουμε την γλώσσα της Κομισιόν γιατί αυτό είναι ένα σημαντικό τμήμα ολόκληρης της αξιολόγησης. Δύο-τρεις γενικότεροι τομείς που τους έχω αναφέρει στο έγγραφο και που σχετίζονται σε θέματα με θέματα με παιδιά, μη συνοδευόμενους ανήλικους και παιδιά που ταξιδεύουν ε, ε, μόνα τους, να δούμε δηλαδή πώς θα δοθεί συνεχής φροντίδα και μέρημνα στα παιδιά κατά τη διάρκεια της ε, σύνταξης ολόκληρης της οδηγίας. Αυτό είναι ένα γενικό, γενικότερο θέμα, ωστόσο σε ένα από τα εκτιμώντας η Κομισιόν έχει πει πιο πολλά πράγματα για το πώς θα πρέπει να πλαισιωθεί το συμφέρον του παιδιού και θα πρέπει ίσως να μας δώσει μια πιο λεπτομερή εξήγηση για το τι σημαίνουν όλα αυτά και το άρθρο θα πρέπει να συμμορφωθεί με το, να, να συμβαδίζει με το εκτιμώντας. Υπάρχουν και θέματα που αφορούν τον ορισμό των μελών της οικογένειας. Η Κομισιόν προτείνει τη συμπερίληψη των έγγαμων ανηλίκων. Ξέρω όμως ότι θα, πρέπει, θα θέλουν να το σκεφτούν οι συνάδελφοι. Και αυτό που έχουμε δει, πρέπει να, μάλλον και αυτό πρέπει να το πράξουμε στο πλαίσιο του συμφέροντος του παιδιού. Το γεγονός ότι ένα παιδί είναι παντρεμένο τον βγάζει από το πεδίο του, του παιδιού και παραμένει μόνο παντρεμένος. Ε, αυτό πρέπει να τα σκεφτούμε. Το φίλο είναι κάτι ακόμα. Η Κομισιόν έχει προτείνει στο άρθρο 10, στο εκτιμάνταση 29, ότι το φύλλο θα πρέπει ρητά να λαμβάνεται υπόψη σε θέματα κοινωνικών ομάδων. Ε, μπορούμε επίσης να μιλήσουμε για την ταυτότητα του φύλλου, για να πώς αφηνήσουμε ότι και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τα αιτήματα προστασίας. Τέλος, το θέμα της ε, πάυσης ενός ειδικού καθεστώτος. Η Κομισιόν προτείνει την προσθήκη μιας ρήτρας ε, ε, που θα συμπεριλαμβάνει επιτακτικούς λόγους για να μην λήξει αυτό το ειδικό καθεστώς. Αλλά υπάρχει και εδώ ένα ερώτημα για το πώς αυτές οι ρήτρες, τι αντίκτυπο μάλλον έχουν αυτές οι ρήτρες στα παιδιά και αν χρειάζεται ειδική αναφορά σε αυτό ή αν η Επιτροπή μας θεωρεί πως ε, το γενικότερο πεδίο της ε, ε, οδηγίας καλύπτει επαρκώς αυτά τα θέματα. Αυτά λοιπόν λέει το έγγραφο εργασία με... Προφανώς τα μέλη της Επιτροπής μπορεί να ανταποκριθούν πολύ διαφορετικά και θα ήθελα πολύ να ακούσω τι έχετε να πείτε και να προχωρήσουμε να δούμε και να εξετάσουμε την έκθεση βέβαια και τις τροπολογίες που μπορεί να φτάσουν σε το χρόνο από τα μέλη. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Lambert. Ευχαριστώ κύριε Λάμπερτ. Να ακούσουμε τώρα τη Βελγική Προεδρία. Αν θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είπατε κι εσείς, Τα θέματα του ασύλου είναι πολύ σημαντικά για την ε, ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου και θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα θέμα στο οποίο πρέπει να προχωρήσουμε και, πάρα πολύ γρήγορα προκειμένου να σεβαστούμε και την προθεσμία του 2012. Να μιλήσω καταρχάς ε, για τα όσα έχει κάνει η κυρία Λάμπερτ. Εξαιρετική δουλειά. Φαίνεται άλλωστε και από το έγγραφο εργασία. Πολλά στοιχεία που αναφέρονται εδώ είναι στοιχεία τα οποία ε, συζητούνται και στο Συμβούλιο. Όσον αφορά τώρα το Συμβούλιο, θα πρέπει να πω ότι είμαστε διατεθειμένοι να ξεκινήσουμε διάλογο το συντομότερο δυνατόν και επομένω με χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο γνωμοδότηση για αυτή την οδηγία και προβλέπεται για την επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής σας. Από πλευρά Συμβουλίου επίσης να σας πω ότι θέλουμε να υποφοληθούμε από τα όσα ετοίμασε η Ισπανική Προεδρία που έχει κάνει μια έξοχη τεχνική προετοιμασία προς το παρόν ε, προχωρούμε τις τεχνικές συζητήσεις ε, προκειμένου να τις ολοκληρώσουμε τις επόμενες εβδομάδες και θα ε, τεθεί υπόψη του Συμβουλίου το κείμενο στις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να ξεκινήσει και ο διάλογος αργότερα. Να πω ότι ο στόχος της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποστηρίζεται από το Συμβούλιο, δηλαδή αυτό που ζητούμε είναι περαιτέρω εναρμόνιση, διασαφήνιση ε, των ορισμών της διεθνούς προστασίας και ταυτόχρονα μία προσέγγιση στο καθεστώς του πρόσφυγα και ε, στο καθεστώς της εμπουκουρικής προστασίας. Τα πάντα είναι σε διαδικασία καθορισμού ακόμα στο Συμβούλιο. Θα είμαστε έτοιμοι σύντομοι και θα το συζητήσουμε στο Συμβούλιο για να ετοιμάσουμε και την άποψή μας. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα, μήπως θέλει να συμμετάσχει στη συζήτηση, ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα για να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Τζιν Λάμπερτ, για το σχέδιο κειμένου που ετοίμασε επισημαίνει τα βασικά στοιχεία και το γενικότερο πνεύμα της πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν έχουμε βέβαια τίποτα το ε, καινοτόμου, αλλά απλώς ε, εκλογικεύουμε και προσπαθούμε να δούμε τα στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να καθορίσουμε κάποιον στο καθεστώς πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, καθώς επίσης να λάβουμε υπόψη και τις πρόσφατες αποφάσεις του δικαστηρίου στο Λουξεμβούργο και στο Στρασβούργο και να έχουμε και προσέγγιση δικαίου για τους ανθρώπους που ζητούν ε, καθεστώς πρόσφυγα και καθεστώς επικουρικής προστασίας. Για να επανέλθω στη χθεσινή συζήτηση, αυτά τα στοιχεία βρίσκονται βρίσκονται και στη συζήτηση για να προσπαθήσουμε να ε, μειώσουμε το χάσμα της αποτελεσματικότητας στα διοικητικά θέματα ε, με στόχο να προσπαθήσουμε να ε, βοηθήσουμε τους ανθρώπους που βρίσκονται στο καθεστώς πρόσφυγα. Όπως είπε η Προεδρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και αυτή υπέρ της επιτάχυνσης των συζητήσεων επί του θέματος και όπως ε, βλέπετε ε, κατέρωθεν υπάρχουν ευνοϊκές συνθήκες προκειμένου να υπάρξει ένας καρποφόρος διάλογος μεταξύ των ε, νομοθετών στις επόμενες εβδομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε λοιπόν τη συζήτηση. Κύριε Ρομέρο Λόπεθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Φρονώ ότι είναι πάρα πολύ καλό το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε προσπάθεια για να βελτιώσει την οδηγία του 2004, διότι έπρεπε να εναρμονιστεί το καθεστώς για να αποφύγουμε και τις καταχρήσεις από πλευράς κρατών μελών όταν εξετάζει ποιοι ε, θα πρέπει να υποφελούνται επικουρικής προστασίας και ποιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο καθεστώς πρόσφυγα. Ε, είναι περίπλοκη νομοθεσία, ε, σχετίζεται πάρα πολύ και με την οδηγία για τις διαδικασίες και νομίζω ότι με τις βάσεις που έχουμε θέσει θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτή την έκθεση. Διότι πράγματι υπάρχουν καταχρήσεις που μπορεί να προκύψουν από τις ε, ε, ελλείψεις που υπάρχουν στους ορισμούς στην πρώτη οδηγία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μελετήσουμε τους πόρους για να δούμε ε, και σε τι υπακούν οι διάφορες αιτήσει που έγιναν. Διότι την τελευταία δεκαετία η μείωση στις αιτήσει ασύλου ήταν σε κάποιες χώρες ε, ακόμα και πονίδιστη θα μπορούσαμε να πούμε. Δεν λειτουργήσε καλά το σύστημα και οι πιέσεις που ασκήθηκαν σε κάποιες χώρες ήταν πάρα πολύ υψηλές. Ίσως δεν ε, δόθηκαν τόσες πολλές εξηγήσει και για το λόγο του τρόπου με τον οποίο ήταν οδηγία, διατυπωμένη η οδηγία και με τον τρόπο όμως με τον οποίο πρέπει να δράσουμε. Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς είναι διαμορφωμένη αυτή η οδηγία και αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό για να επιμείνουμε στις αιτήσει που έχουν γίνει και για να μειώσουμε όλα αυτά τα κενά τα οποία όπως είπε η συγγήτρια εξακολουθούν να υφίστανται. Όλα όσον αφορά τα θέματα προστασίας, τα μέλη της οικογένειας, τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Μία σειρά δηλαδή ε, από στοιχεία που δημιουργούν ένα νέο καθεστώς που δεν ε, συμβιβάζεται με τα όσα λέει η Γενέβη και σαφώς θα πρέπει να τα βελτιώσουμε για να μην ε, δώσουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να έχουν αμφίσιμες θέσεις. Και επίσης να μην δικαιολογείται αυτή η τεράστια μίαση που είχαμε στις αιτήσεις ασύλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χολμάγερ. Ναι, Πρόεδρε, αγαπητέ συνάδελφοι, να ευχαριστήσω την Τζιν Λάμπερτ για το εξαιρετικό έγγραφο και για την προθυμία με την οποία συνεργάστηκε μαζί μας ε, για την ε, αναγνώριση της οδηγίας για τις ε, δεξιότητες. Σε κάποιους τομείς βλέπω ότι έχουμε κοινέ θέσεις. Το ερώτημά μου έχει να κάνει και με την εξέταση στο, της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί ε, στις διάφορες χώρες ε, για τα ίσα δικαιώματα, για, για την ε, εξίσωση μάλλον προσφύγων και των όσων βρίσκονται στην χώρα. τι γίνεται με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ας πούμε. Τι γίνεται με τις γενικές κοινωνικές πρόνοιες που δίνει στους ανθρώπους αυτούς η κάθε χώρα. Γιατί όντω ε, δημιουργούνται προβλήματα όταν υπάρχει τέτοια είδου εξίσωση, ε, ευτυχώ ή δυστυχώ, στα κράτη-μέλη. Υπάρχει δηλαδή μεγάλη αντίσταση από τα κράτη-μέλη να δεχτούν ω ίσου του πρόσφυγε. Δεύτερον, άλλο ένα δύσκολο θέμα για το ποιο παρέχει την προστασία. Θεωρώ πολύ σωστό ότι όντω θα πρέπει να κάνουμε μία ανάλυση για το κατά πόσο είναι ε, σωστό ε, να υπάρχει και μια εναλλακτική λύση σε κάθε κράτος μέλος. Για αυτούς δηλαδή που έρχονται να ζητήσουν άσυλο και να παραμείνουν στις χώρες μας. Ε, γιατί υπάρχουν πολλές χώρες στις, στον κόσμο που δεν είναι οι μόνο οι κρατικές αρχές που δίνουν την προστασία, που παρέχουν την προστασία στους πρόσφυγες, υπάρχουν και άλλοι φορείς. Οπότε ίσως να έπρεπε και εμείς να συμπεριλάβουμε ένα βαθμό ευελιξίας σε, αυτή την, σε αυτό το έγγραφο. Επίσης, τα μέλη των οικογενειών η, η, ο όρος οικογένεια ορίζεται σαφώς στην οδηγία για τις α, ε, δεξιότητες και αυτό ίσως να είναι λίγο προβληματικό, ειδικά με τις, σε ό,τι αφορά τις ε, α, με το Συμβούλιο. Γιατί νομίζω ότι η, διεύρυνση του όρου οικογένεια θα οδηγήσει στο εξή. Θα, υπάρξει, ε, θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα, θα υπάρξει παραβίαση της, του όρου αυτού Η διεύρυνση λοιπόν του όρου όντως ε, προσκρούει σε προβλήματα. Θα μπορούσαμε εδώ πέρα να θέσουμε μεγάλες απαιτήσει, αλλά αν δεν υπάρχει καμία συμφωνία με το Συμβούλιο, ε, τότε θα είναι προβληματικό. Γιατί η δική μας ε, θέση προφανώς είναι να πάμε λίγο προς τα μπρος, να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα από τα βασικότερα προβλήματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε με το Συμβούλιο. Και θα πρέπει να το δούμε. Τώρα, το θέμα των ψυχικών ασθενειών και της παροχής βοήθειας στα άτομα που τη χρειάζονται. Ε, το θέμα αυτό έχει οριστεί, δηλαδή ξέρουμε τι σημαίνει ακριβώς ψυχικό πρόβλημα. Γιατί και με ψυχολόγους να συζητήσετε είναι πολύ ευρύς όρος αυτός. Μπορεί να είναι διάφορα πράγματα το πρόβλημα το ψυχικό ή μπορεί να, είναι, να προκύπτει και από διάφορους, ε, και για διάφορους λόγους. Ε, γιατί κάποιος έχει ας πούμε ένα ψυχικό τραύμα από την παιδική του ηλικία στην χώρα του, γιατί δεν μπορεί να προσαρμοστεί στη νέα κοινωνία που βρίσκει. Ε, είναι λοιπόν πολύ δύσκολο το θέμα αυτό. Μάλλον λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε αφού είναι δύσκολο και να το ορίσουμε. Μήπως θα πρέπει να συζητήσουμε αν γενικώ για τα άτομα με ψυχικά προβλήματα πρέπει να δοθεί ένα ιδιαίτερο καθεστώς. Και επίσης, αν κάποιος δεν διώκεται στη χώρα του, αλλά έχει, ε, προσπαθεί να βγει από τη χώρα του ή αν έχει ε, ψυχικά προβλήματα. Τι σημαίνει ότι δεν μπορεί να ζήσει στη χώρα του. Δηλαδή, εμείς πρέπει ε, κάποιον να, τον, να το στείλουμε πίσω στην χώρα του. έχει, δεν έχει ψυχικά προβλήματα μόνο και μόνο επειδή δεν διώκεται εκεί μήπως αυτά πρέπει λίγο να τα δούμε περισσότερο. Και αυτό ειδικά με τα ψυχικά προβλήματα πρέπει νομίζω να το συζητήσουμε εντελεχέστερα. Τώρα, τους, ε, για τους ε, ύπανδρους ανήλικους. οι συνήθως αυτοί είναι, έχουν υποχρεωθεί να παντρευτούν, οπότε δεν έχουν ιδιαίτερη δυνατότητα να πούνε ή να δηλώσουν ότι υποχρεωτικά αναγκάστηκαν να παντρευτούν, ότι τους πάντρεψαν. Νομίζω η Κομισιόν δεν θέλει να ασχοληθεί τόσο πολύ με το θέμα των υποχρεωτικών ε, γάμων, των αναγκαστικών γάμων. Αυτό βέβαια εμπίπτει και στο θέμα των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν κάποιο είναι 17 χρονών και θέλει να παντρευτεί το φίλο του ή τη φίλη του και έχει την, ε, την, είναι δική του η απόφαση, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι... Στις ε, περισσότερες ε, περιπτώσεις δεν συμβαίνει αυτό. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να επιλέξουμε έναν διαφορετικό, μια διαφορετική άγουσα. Και επίσης τα, τα θέματα εκπαίδευση των παιδιών, πρόσβαση στα σχολεία. Φυσικά τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση. Είτε πρόκειται να επιστρέψουν στα πατρίδα του, είτε θα μείνουν στι δικέ μα χώρε. όπου και να ζήσουν πρέπει να έχουν πρόσβαση σε σχολείο, σε εκπαίδευση για τις δυνατότητες ένταξης ε, και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Σωστό είναι που λέμε ότι πρέπει να υπάρξει ένταξη ε, για αυτούς που θα παραμείνουν στις χώρες μας, αλλά αν δούμε την όλη οδηγία και θέλουμε να έχουμε μια σύντομη και συνεκτική διαδικασία που θα κρατήσει ας πούμε έξι μήνες και θα τελειώσει, τότε είναι δύσκολο μέσα αυτούς τους έξι μήνες να δώσουμε ιδιαίτερες προσφορές στα παιδιά, να τους δώσουμε ε, δυνατότητες εκπαίδευσης, γιατί σε 3 μήνες ας πούμε από την ώρα που θα τους, θα τους δώσουμε τις επιλογές αυτές θα πρέπει να φύγουν και να γυρίσουν πίσω στις χώρες τους για, τους, για όσους θα παραμείνουν στις χώρες μας φυσικά ε, είναι σημαντικό και είναι ε, εκ των όνων να τους προσφέρεται πρόσβαση στην ε, εκπαίδευση. Βεβαίως εδώ υπάρχει και συνευθύνη αυτού που μένει στη χώρα. Αυτού που θέλει να μείνει στη δική μας τη χώρα. Δηλαδή θα πρέπει και οι άνθρωποι αυτοί να προσπαθήσουν να ενταχθούν, όχι να περιμένουν μόνο να τους εντάξει κάποιος. Αυτοί που παραμένουν στις δικές μας χώρες πρέπει να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν ότι και να το πούν ότι θέλουν να ενταχτούν, θέλουν να μάθουν τη γλώσσα της χώρας που μένουν ή που θέλουν, στην οποία θέλουν να ενταχτούν και ότι δεν υπάρχει απλώς μία ευθύνη, ε, ούτε είναι χρέος της χώρας να τους εντάξει. Οι ίδιοι θέλουν να ενταχτούν, οπότε θα πρέπει να κάνουν και αυτοί μια σοβαρή προσπάθεια. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στο συμφέρον των παιδιών. Είναι πολύ σημαντική αυτή η παρατήρηση, διότι πλέον βάσει της συνθήκης της Λισιφοβόνας ε, ισχύει ε, αυτό και μπορούμε να ε, υψώσουμε τον πύχη, διότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας και χρειάζονται επιπλέον φροντίδα. Δεν αρκεί κατ' με να αναφερθεί κάτι τέτοιο σε μια αιτιολογική σκέψη. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Τι σημαίνει στην πράξη για το κράτος μέλος. Θα πρέπει να υπάρχει στο διατακτικό, σε ένα άρθρο. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπρόνς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες προσφύγων. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι έχουν εντοπιστεί ε, προσωπικά και διώκονται από το κράτος μέλος ε, και δεύτερον υπάρχουν αυτοί οι οποίοι απλώς φεύγουν από επικίνδυνες χώρες. Οι πρώτοι μπορεί να είναι κάλλιστα πρόσφυγες αρκεί να μην έχουν παρακάμψει ε, ασφαλείς χώρες. Οι δεύτεροι έχουν τη συμπάθειά μας, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε όλο τον πληθυσμό καταπιεσμένων χωρών όπως είναι η Κίνα, το Αφγανιστάν και άλλων αφρικανικών χωρών. Θα ήταν αδύνατον. Ακόμα και αν τους δεχόμασταν, γιατί θα έπρεπε να αφήσουμε τον υπόλοιπο πληθυσμό να ζει στη χώρα. Μήπως δεν θα έπρεπε να καλέσουμε όλη την Κίνα, όλο το Αφγανιστάν, ε, αν είναι να είμαστε συνεπείς σε αυτά που κάνουμε. Δεύτερον, επικρίνουμε πολλές χώρες γιατί δεν ανοίγουν τις πόρτες τους σε όλο και περισσότερους πρόσφυγες, αλλά αν δείτε τις ε, δημοσκοπήσεις, ε, οι κάτοικοι των χωρών ζητούν να αναλυφθεί δράση ώστε να σταματήσει αυτή η ροή. Δηλαδή το αντίθετο ακριβώς. Ορισμένε φορές αυτά που κάνουμε φαίνονται πολύ ευγενικά. Ε, λέμε ότι θα πρέπει να δοθεί μια θέση εργασίας ή ένα σπίτι σε ένα πρόσφυγα κατά προτίμηση σε ένα κράτος μέλος. Ουσιαστικά λέμε ότι ο πολίτης της χώρας μέλο δεν θα πρέπει να λάβει θέση εργασίας ή σπίτι και να το πάρει ο πρόσφυγα. Κάποιοι από αυτούς που έχουν φύγει από επικίνδυνες χώρες το έχουν κάνει γιατί έχει δράσει κατά συγκεκριμένο τρόπο ε, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς ακόμα και η δική μου ξεκίνησε πόλεμο κατά του Ιράκ. Ε, εάν σταματήσουμε να ξεκινούμε τέτοιες δράσεις, τέτοιες διενέξεις, ίσως να είναι πιο ασφαλείς οι χώρες ε, που, που ζουν οι άνθρωποι αυτοί. Κάποιες φορές ε, έχουμε πρόσφυγες οι οποίοι φεύγουν ε, γιατί διώκονται λόγω καταπιεστικών ε, νόμων που δεν τους επιτρέπουν την ελευθερία του λόγου. Κατανοούμε βέβαια όλους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πάρα πολλές χώρες αυτές που έχουν ελευθερία του λόγου, αλλά φαντάζομαι ότι εάν διώκονται στη χώρα τους για αδικήματα που διέπραξαν στη χώρα τους, θα συλληφθούν ούτως ή βάσει του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και θα επιστραφούν στη χώρα τους. Ευχαριστώ βλέπω ε, κάποιον άλλο να θέλει το λόγο. Να ζητήσω από την εισηγήτρια λοιπόν, ε, την κυρία Λάμπερτ, να ε, ολοκληρώσει τη συζήτηση Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συνεισφορά τους. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε λίγο περαιτέρω. Κάποια πράγματα βέβαια έχουν σχέση και με την οδηγία για τις διαδικασίες, ε, το να φροντίσουμε δηλαδή κάθε υπόθεση να εξετάζεται αυτόνομα. Το να συμπεριληφθεί βέβαια κάτι στο κείμενο τη οδηγία δεν σημαίνει ότι όποιο έχει προβλήματα ψυχική υγεία ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με καταναγκαστικού γάμου ή οτιδήποτε άλλο δεν θα εξετάζεται αυτόνομα και θα βρίσκονται στο καθεστώ προστασία. Γι' αυτό ακριβώ εξετάζουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά και αξιολογείται η κάθε περίπτωση και ε, εξετάζουμε τι κίνδυνος υπάρχει αν επιστραφεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος στη χώρα του. Μας ενδιαφέρει ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διαδικασίες. Ξέρω ότι κάποιες χώρες έχουν πολλά προγράμματα με το UNHCR για να δούνε πώς εφαρμόζονται τα διάφορα προγράμματα, κάτι το οποίο κατά μένα είναι πολύ σημαντικό, διότι η νομοθετική πλευρά δεν λύνει όλα τα προβλήματα. Μας δίνει το πλαίσιο, αλλά δεν μας ε, λύνει όλα τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε σε κάθε περίπτωση. Ένα από τα θέματα το οποίο αναφέρθηκε ως ερώτημα και ίσω θα μπορούσαμε να επανέλθουμε σε αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το θέμα των εφήμων και τι γίνεται όταν κάποιος είναι αντίθετο σε ένα συγκεκριμένο έθιμα το οποίο θεωρούν ότι τους καταπιέζει και κατά πόσον αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην αξιολόγηση, κατά πόσον το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούν ότι καλύπτεται επαρκώς αυτό στο κείμενο ή θεωρείται ε, ως πολιτικό δικαίωμα για να μπορεί κάποιος να πει την άποψή του ή θεωρείται καταπίεση. Μήπως αυτό εντάσσεται σε κάποια άλλη κατηγορία. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί και να εξεταστεί περαιτέρω. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, κυρίως για το, ε, την πρόσπιση των συμφερόντων των παιδιών. Τα θέματα της προστασίας είναι το ένα τμήμα, το ένα σκέλος ε, των διεθνών εξελίξεων. Υπάρχουν θέματα ανάπτυξης, θέματα εμπορίου, τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Το θέμα της αγοράς εργασίας νομίζω ότι έχουμε τρία κρατημέλη αυτή τη στιγμή που έχουν διαφορές σε θέματα πρόσβασης ε, με την, ε, στην αγορά εργασίας και με τις τρεις κατηγορίες Νομίζω ότι κανένας δεν θα θεωρήσει ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός θέσεων εργασία σε μία αγορά εργασίας. Το πώς ε, λοιπόν ο καθένα ε, θεωρεί ότι ταιριάζει με την αγορά εργασία τους και αν υπάρχουν τέτοιε δυνατότητε, δεν είναι θέμα προγράμματος, είναι θέμα του πώς ε, είναι οι συγκυρίε εποχές. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να το παρουσιάσουμε ως κάτι σταθερό ότι έχουμε ξέρω εγώ χι εργασίας και αν πάρεις μία κάποιο θα, χάσει τη θέση του ε, θα πρέπει να δούμε πώς έχει αγορά εργασίας η οικονομική κατάσταση και το σύστημα ένταξης και ασφάλειας για τον καθένα ε, αυτό όμως είναι μάλλον αρμοδιότητα άλλων επιτροπών και όχι της δικής μας όπως είπα λοιπόν και πάλι, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Πολλά από αυτά θα συμπεριληφθούν στην πρόταση έκθεσης που θα κάνω, αλλά είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε και τροπολογίες και από τους υπολείπους και προσβλέπω στη συζήτηση και τη συνεργασία και όταν θα έχουμε εμείς διευκρινίσουμε ποια είναι η δική μας η θέση, τότε νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε και πολύ επικοδομητικές συζητήσεις με τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λάμπερτ αν κατάλαβα καλά δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε από την Προεδρία. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστούμε όλους όσους ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Να προχωρήσουμε τώρα στο επόμενο σημείο, 16. Και πάλι, τροποποίηση του κανονισμού 539-2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών. Διακόπτη πρόεδρος. Αχ, συγγνώμη, ξεχάσαμε το 15. Έχουμε και ένα σημείο πριν. Στο 15 λοιπόν, επέκταση του πεδίου εφαρμογή της οδηγίας στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Εισηγητής ο κύριος Μωράες. για να δούμε το σχέδιο έκθεσης και να δούμε πώς έχει κατάσταση. Έχουμε επίσης ε, ε, παρουσία της Βελγικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς όμως να ακούσουμε την έκθεση του εισηγητή του κυρίου Μωράς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Αυτό το θέμα στην προηγούμενη θητεία το είχε αναλάβει η συνάδελφος ε, Ρουρ, αλλά δεν μπόρεσε να βρει συμφωνία πριν να αρχίσει να ισχύει η Λισαβόνα. Και τώρα έχουμε μια ευκαιρία να προχωρήσουμε στο πλαίσιο της Βελγικής Προεδρίας για μια πρόταση που πιστεύω ότι έπρεπε εδώ και πολύ καιρό να έχει περάσει για να μπορέσουν να ωφεληθούν όλοι όσοι χρειάζονται διεθνή προστασία Σύντομα, να σας πω την γενική μου προσέγγιση. Υπάρχουν τρεις τομείς όπου εγώ αποκλίνω από τις προτάσεις του Συμβουλίου. Να προσθέσω ότι στις 7 Σεπτεμβρίου στην συνάντηση των σκιωδών εισηγητών είχαμε μια εξαιρετικά επικοδομητική ε, συνάντηση με όλες τις πολιτικές ομάδες ήμασταν σύμφωνοι, γι' αυτό και δεν διαβλέπω προβλήματα. Να υπογραμμίσω τρία σημαντικά σημεία. Καταρχήν, όπως σας είπα, έχουμε φτάσει μια... ελπίζω ότι θα έχουμε μια ε, συμφωνία με το Συμβούλιο μας τα Χριστούγεννα και γι' αυτό η προσέγγιση που θα ακολουθήσω είναι να ε, λάβω υπόψη τις περισσότερες προπιθανές τροπολογίες της Κομισιόν τρεις ε, κεντρικοί τομείς όπου αποκλίνω από το του συμβιβαστικό κείμενο του Συμβουλίου είναι καταρχήν θέλω να στηρίξω την πρόταση της Κομισιόν ότι πλήρης διάρκεια της διαδικασίας ασύλου να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των πέντε ετών για την νόμιμη παραμονή Έπειτα η απέλαση να είναι μόνο πιθανή στο πρώτο κράτος μέλος και όχι σε μια τρίτη χώρα, γιατί εκείνοι φέρουν την πλήρη ευθύνη για την ε, απέλαση καθώς έχουν όλες τις πληροφορίες για τον πρόσφυγα και την κατάστασή του. Τέλος, να εξασφαλίσω ότι η αρχή της ε, ενότητας της οικογένειας θα στηριχθεί. Το Συμβούλιο βασικά συμφωνεί, αλλά υπάρχουν κάποια σημεία που αφορούν την διατύπωση και ε, στην η κυρία Σαργεντίνη στη συνάντηση των σχεδόν εισηγητών έθιξε το, γεγον... το θέμα του αν ένα μέλος της οικογένειας είναι υποχρεωμένο ή όχι να ακολουθήσει έναν ε, πρόσφυγα που απελάβνεται. Γενικά ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να αποκλείει την είσοδο των μελών της οικογένειας. Μπορεί μια οικογένεια να μην θέλει να ακολουθήσει τον πρόσφυγα. Μπορεί να υπάρξουν τέτοιες ε, περιπτώσεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει η διατύπωση να είναι πιο ακριβής και τελικά οι αρισκαιώτες είναι όλοι ικανοποιημένοι με τη τελική διατύπωση. Χρονοδιάγραμμα, όπως σας είπα, είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση στις 7 Σεπτεμβρίου. Επόμενη συνάντηση των θα είναι 6 Οκτωβρίου και ο πρώτος τριμερής διάλογος στις 12 Οκτωβρίου. Και πάλι να τονίσω ότι θέλουμε να φτάσουμε σε συμφωνία υπό την Βελγική ε, Προεδρία. Και αισιοδοξώ πως θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ κύριε Μωράης. Η Βελγική Προεδρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήθελα κυρίως να μιλήσω για τη συνεργασία μας στους άλλους φακέλους ε, για το άσυλο. Δηλαδή θα κάνω μια πρώτη εισαγωγή και μετά θα επανέλθω στο θέμα αυτό θα πρέπει να δούμε τι γίνεται στο Συμβούλιο. Όπως είπα, το άσυλο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης του Συμβουλίου των Υπουργών τον Ιούλιο, παρουσίασε μια στρατηγική πρόταση που περιείχε τους στρατηγικούς στόχους για το 2012 για το σύστημα ασύλου. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ήδη προέβλεπε μια στρατηγική και για την καλύτερη επίτευξη των στόχων αυτών αυτή η στρατηγική υποστηρίχτηκε και από τους υπουργούς. Σημαίνει αυτό ότι είναι δυνατόν να γίνουν πρόοδοι σε σύντομες ε, προθεσμίες. Θα πρέπει δηλαδή ε, να δοθεί μια κάποια δυναμική, μια κάποια όθηση για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το σύστημα του ασύλου μέσα στο 2012. Ε, Μπορούμε βέβαια να συζητήσουμε και για τις ε, διαδικασίες. Αλλά η φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε με όλα τα κείμενα. Με... Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, σε μια πρώτη βάση θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ε, συμβαστικές, γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η δυναμική, υπάρχει αυτή η όθηση και μπορεί έτσι να δοθεί μια ε, μεγαλύτερη δυναμική και στα υπόλοιπα κείμενα του, του ασύλου. Επίσης θα πρέπει να δούμε πού έχουμε πιθανότητες να ολοκληρώσουμε σύντομα. Για το 2012 Έχουμε να πούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σύντομα και όλοι οι φορείς και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν παρόντα για τη συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου ε, στην ε, Κορεπέρ. Είχαμε πολύ χρήσιμες συζητήσεις εκεί. Αλλά για να επανέλθουμε τώρα στο συγκεκριμένο ζήτημα, ένα από τα θέματα προτεραιότητας, δηλαδή οι μακροχρόνοι κάτοικοι, οι... εμείς θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Μωράης για τη δουλειά που έκανε Καταρχήν, στην προετοιμασία αυτής της έκθεσης, όπως είπε και ο ίδιος, Υπήρχε σαφής βούληση από πλευράς όλων των θεσμικών οργάνων να σημειωθεί πρόοδος εδώ και γι' αυτό και θέλω να σας ευχαριστήσω και για την αισιοδοξία σας ε, σαφώς υπάρχει βούληση να προχωρήσουμε γρήγορα σε συμφωνία και πιστεύουμε πως είναι σημαντική μια γρήγορη συμφωνία γιατί είναι ένα κείμενο το οποίο είναι επιτάπητο στο Συμβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πριν να ξεκινήσει η Λισαβόνα δεν, μπόρεσε να βρούμε, δεν μπορέσαμε να βρούμε συμφωνία όμως νομίζω πως τώρα θα πρέπει να, κάνουμε, να φτάσουμε σε μια συμφωνία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Υπήρχε βέβαια η συμβιβαστική του Συμβουλίου που ολοκληρώθηκε το 2008 που σχεδόν είχαμε ομοφωνία. Και αυτό μας έβαλε ως Προεδρία σε πολύ ευνοϊκή θέση, γιατί είχαμε μια σαφή θέση του Συμβουλίου. Ο κύριος ε, Μωράης και το σχέδιο έκθεσής του υποβλήθηκε στις αρμόδιες αρχές στο Συμβούλιο και από αυτές τις βάσεις θα αναπτύξουμε και την θέση του Συμβουλίου. Πιστεύουμε πως το σχέδιο έκθεση είναι καλή βάση συμβιβαστική γιατί όπως είπε ο κύριος Μωράης ήδη πολλές από τις αλλαγές που είχαν γίνει στο Συμβούλιο, στην πρόταση της Κομισιόν, έγιναν, είχαν γίνει δεκτές και στο κείμενό του, έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενό του. Υπάρχει λοιπόν βάση για συμφωνία, υπάρχουν κάποια σημεία ωστόσο που υπάρχουν, ε, ε, συνεχίζουν να ε, υπάρχουν αποκλήσεις, αλλά ελπίζω πως σύντομα το είπατε και εσείς στις 12 Οκτωβρίου, θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε διάλογο για όλα αυτά. Σκοπεύουμε να μπούμε σύντομα σε διάλογο και με τα άλλα θεσμικά όργανα και με τη βάση της έκθεσης του σχεδίου άλλων έκθεσης τη κυρίας Λάμπρεχ θα ε, καταλήξουμε και εμείς σε μια θέση για το Δουβλίνο. Ε, αυτό είναι επιτάπητος εδώ και χρόνια. Ε, τεχνική δουλειά έχει γίνει υπό την Τσεχική και τη Σουηδική Προεδρία και εμείς βασιζόμαστε σε αυτήν τη δουλειά που έχει ήδη ολοκληρωθεί. Και μέσω πρόθεσμα ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε τις τεχνικές αυτές συζητήσεις και να καθορίσουμε τη θέση μας, καθώς και να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τα θεσμικά όργανα και τους εισηγητές. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια έκθεση για πρώτη ανάγνωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δική σας θέση λοιπόν είναι ξεκάθαρη επί τη βάση αυτής της έκθεσης και φιλοδοξούμε να καθορίσουμε τη θέση του Συμβουλίου και να ξεκινήσουμε διάλογο σύντομα. Βέβαια, από πολιτική άποψη είναι πολύ ευαίσθητο αυτό το θέμα. Και υπάρχουν κάποια σημεία όπου οι προτάσεις ξεπερνούν το πεδίο του μέσου. Για το Eurodac. Περιμένουμε νέα πρόταση της Κομισιόν που ελπίζουμε ότι θα κατατεθεί σύντομα. Επί τη βάση προηγούμενων προτάσεων έχουμε λίγο πολύ καταλήξει, ολοκληρώσει μάλλον τις συζητήσεις στο Συμβούλιο και έχουμε θέση. Επ' αυτού το Κοινοβούλιο επίσης έχει υιοθετήσει θέση και νομίζω ότι επί τη βάση προηγούμενων συζητήσεων μπορούμε να καταλήξουμε ότι σε μεγάλο βαθμό σκεφτόμαστε περίπου τα ίδια. Ελπίζω πως και εδώ θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Όπως είπα, οι όροι προστασίας δεν έχουν αγνοηθεί. Έχουμε συζητήσει την οδηγία περί διαδικασίας εδώ εχθές και στο Συμβούλιο συνεχίζουμε τις τεχνικές συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Είναι φυσικά ζητήματα που από πολιτικής άποψης είναι πολύ πιο δύσκολα και λεπτά συνεχίζουμε τις εργασίες σε τεχνικό επίπεδο και χρησιμοποιούμε την υπουργική διάσκεψη στις αρχές του μήνα ώστε να το δούμε αυτό από πολιτικής άποψης και να δούμε δηλαδή να σφιγμομετρήσουμε τον αντίκτυπο των προτάσεων της Κομισιόν και όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο γύρος συζητήσεων θα έχουμε μια θέση για την έκθεση της κυρίας Γκυγιόμ που στη συνέχεια θα μας βοηθήσει να καθορίσουμε τη στρατηγική μας και να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας για κοινό σύστημα ασύλου μέχρι το 2012. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ τώρα η κυρία η Κομισιόν, η κυρία Γκάλ. Ναι, για την οδηγία για τους ε, μακροχρόνους ε, ε, κατοίκους Νομίζω πω η έκθεση του κ. Μωράη αποτελεί μια εξαιρετική βάση κίνησης για ταχύε διαπραγματεύσεις στους επόμενες εβδομάδες. Εγώ πιστεύω πως ένα από τα σημεία κλειδιά των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στους συν θα είναι πιθανότατα η μέθοδος υπολογισμού της περίοδου αναμονής για να πάρει κανείς το καθεστώς Όπω το είπα και στον εισηγητή και στου σκιώδε στι αρχέ του Σεπτεμβρίου, η Κομισιόν μπορούσε να στηρίξει τη συμβεβαστική του Συμβουλίου, που επετεύχθη στο τέλο του 2007 σχεδόν με ομοφωνία, αλλά φυσικά σημειώνουμε πως ο εισηγητή προτείνει για το συγκεκριμένο σημείο να στηρίξουμε την πρόταση της Κομισιόν. Προσπαθούμε πάντως να διευκολύνουμε μια συμφωνία ανάμεσα στους συνομοθέτες και για αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Merci, Madame σας ευχαριστούμε κύριε Γκάλ και θα δώσουμε λοιπόν το λόγο τώρα σε όποιον θέλει. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για το ανοιχτό του πνεύμα και τη συνεργασία του με τους κοιόδους αλλά και με τα άλλα θεσμικά όργανα. Όπως αναφέρθηκε η συνεδρίαση της 7 η Σεπτεμβρίου ήταν εξαιρετικά καρποφόρο και βλέπουμε το αποτέλεσμα με το σχέδιο έκθεσης που μας υποβλήθη. Πόσο σημαντικό ήταν να δούμε σε αυτήν την έκθεση ότι από τη μια πλευρά οι προτάσεις που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που χρονολογούνται από τις 23 Απριλίου 2008 έχουν ληφθεί υπόψη, υπάρχει μια συνέχεια και από την άλλη πλευρά βλέπουμε πως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν ενσωματωθεί και ταυτόχρονα κάποια σημεία εξαιρετικά λεπτά, τα οποία διεκδικούν τα κρατημέλη, προσεκίζονται με μεγάλη λεπτότητα και πάντοτε αυτό το ανοιχτό πνεύμα για διάλογο εν ώψη της προετοιμασίας και του χρονοδιαγράμματος ε, μέχρι το τέλη της χρονιάς. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω μόνο κάποια σχόλια, να επιμείνω για τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν, ότι δηλαδή το σχέδιο της έκθεσης είναι ε, ισορροπημένο, δεν ε, ξεχνά κανένα κεντρικό σημείο και κυρίως την υπεράσπιση των συμφερόντων των δικαιούχων της διεθνούς προστασίας πριν και μετά την χορήγηση αυτού του καθεστώτος ε, ε, Έχουμε δύο παρατηρήσεις πριν από το χορήγηση και δύο μετά. Και αυτό για να ε, διαχωρίσω την, και να εξηγήσω τη θέση μου και να επιστήσω την προσοχή σε ορισμένες διαφορές. Καταρχήν πριν από τη χορήγηση αυτού του καθεστώτος νομίζω πως όλοι συμφωνούμε ότι είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη όταν πρέπει να αποφασίσουν για την απόδοση ή όχι, τη χορήγηση ή όχι του καθεστώτος μακροχρόνιου κατοίκου να λάβουν υπόψη τα περίπτωση ε, τα στοιχεία και την απόφαση να τη λάβουν χωριστά και εδώ συμφωνώ με τη θέση του εισηγητή. Αντίθετα, όπως είπε η Κομισιόν, ένα από τα κεντρικά σημεία είναι ακριβώς ο υπολογισμός των πέντε ετών διαμονής. Βλέπουμε ότι στην έκθεση η πρόταση της Κομισιόν γίνεται ε, δεκτεί και τώρα περιμένουμε τη θέση του Συμβουλίου. Να δούμε αν θα είναι τουλάχιστον το μισό, πώς θα υπολογιστεί. Νομίζω πως είναι ένα κεντρικό σημείο για την έκθεση και από αυτού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση του κ. Μωράης έχει σαφώς εκφράσει την θέση του. Ελπίζω λοιπόν πως οι διαπραγματεύσεις θα είναι καρποφόρες και θα μπορέσουμε να βρούμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Δύο ακόμα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Από τη μια πλευρά, την απόφαση απομάκρυσης από το δεύτερο κράτος μέλος που για μας είναι πολύ σημαντική. Να επισήσω την προσοχή στο γεγονός ότι το Συμβούλιο είχε ζητήσει μια προθεσμία δύο μηνών και στην έκθεση αυτό αναφέρεται, παραμένει μία από τις θέσεις που σαφώς ε, εκφράζει το Κοινοβούλιο. Τέλος, το τελευταίο σημείο ε, ενίσχυση των ενισχύσεων κατά της ε, ε, επαναπροώθησης. Μεταφορά της προστασίας κυρίως όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας και εδώ επιμείνω για τον σεβασμό της επέκτασης του σημερινού πεδίου εφαρμογής της οδηγίας καθώς επίσης και το σεβασμό των εθνικών νομοθετικών διατάξεων και των ευρωπαϊκών νομοθετικών διατάξεων όσον αφορά τα μέλη της οικογένειας. Επ' αυτού λοιπόν δέχομαι όπως είπε και το Συμβούλιο ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω πως στη νέα διαδικασία θα βρούμε μια συμφωνία πάνω σε αυτά τα σημεία. Ελπίζω πως θα γίνει σεβαστό το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος της χρονιάς και να επιταχυνθούν οι διαπραγματεύσεις και έπειτα έχω την εντύπωση πως είναι σημαντικό να προχωρήσουμε ακόμα και αν ο καθένας επιμένει ότι είναι όντως πολύ λεπτό το ζήτημα από πολιτικής άποψης. Σας ευχαριστώ. Mrs. Argentini. κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μωράρας, για τα πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έκανε σε αυτό το έγγραφο. Έχω κάποια σχόλια, αλλά δεν είναι σχόλια επί της πρότασής του. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα της συζήτησης των πέντε ετών πριν ε, δοθεί το καθεστώς. Νομίζω ότι το Συμβούλιο πρέπει να κάνει κάτι από αυτού. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο συμφωνούν από αυτό είναι πολύ περίεργο να κάνουμε εμπόριο ανθρώπων με αυτόν τον τρόπο. Αν κάποιο έχει χρειαστεί να φύγει από τη χώρα του και κάνει αίτηση για το καθεστώ του πρόσφυγα, αυτά τα πέντε χρόνια θα πρέπει να αρχίσουν να μετρούν ματιαφήξει του, διότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό ο άνθρωπο να έχει το δικαίωμα να ξεκινήσει τη ζωή του. Ε, δεν ξέρω αν είπε η περίοδος ε, πέντε ετών ισχύει, ε, μπορεί να έχουν περάσει δύο χρόνια χωρίς να έχει γίνει τίποτα ουσιαστικά έχουμε διαφορετική μεταχείριση υπηκών τρίτων χωρών ανάλογα με την έγκριση που έχουν λάβει. Ο κύριος Μωράες αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό και νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Θα πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα ανεξάρτητης κατοικίας. Μπορεί κάποιος να ξεκινά ως μέλος μιας οικογένειας και μπορεί ο ένας εκ των μελών της οικογένειας να δικαιούται διεθνούς προστασίας και αυτό μπορεί να συνεχιστεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Αλλά αν κάποιο θέλει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, δεν μπορεί να εξαρτάται για όλη του τη ζωή από την άδεια παραμονής κάποιου άλλου. Επομένως, εάν κάποιος έχει προ καθεστώς ε, νομικής προστασίας και εάν ε, κάποιος μεταφερθεί από τη μία χώρα στην άλλη. Τι γίνεται με τα μέλη της οικογένειας. Εάν το επιθυμούν σαφώς πρέπει να πάνε, αλλά αν ε, δεν θέλουν να μεταβούν στη χώρα αυτή, επειδή έχουν διαμείνει ε, σε συγκεκριμένη χώρα για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να ζητήσουν να παραμείνουν. Νομίζω στη χώρα μου μπορεί να γίνει για τρία χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να συγχαρώ τον κύριο Μωράες για την εξαιρετική του δουλειά, η οποία ήταν και ταχύτατα, πάντα σε πολύ καλή συνεργασία με τους κοιόδης εισηγητές, λαμβάνοντας πάντα υπόψη και τις θέσεις μας. Χαίρομαι που ο κύριος Μωράες υποστηρίζει τα πέντε αυτά χρόνια να βασίζονται στη συνεχή διαμονή σε ένα κράτος μέλους και να ξεκινούν όταν το ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάνει πρώτη φορά αίτηση για καθεστώς προστασίας. Θεωρώ ότι φροντίζουμε και τα κράτη-μέλη σε αυτή την περίπτωση. Αυτός ο οποίος ε, έχει καθεστώς ε, μακρά διαμένοντος μπορεί να μεταβεί από τη μία χώρα στην άλλη. Επίσης, Εάν πρόκειται για απέλαση, η απέλαση θα πρέπει να γίνεται μόνο στο κράτος μέλος το οποίο του έδωσε το καθεστώς της προστασίας. Συμφωνώ με αυτό, αλλά λέει ότι τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να απελάσσονται μαζί με αυτόν ο οποίος απολαμβάνει καθεστώς ε, προστασίας. Δεν συμφωνώ με αυτό είναι απαραίτητο σε όλες τις εκθέσεις που έχουμε για, την, για το άσυλο και τη μετανάστευση να έχουμε κατά νου την ε, ενότητα μιας οικογένειας, αλλά επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η ενότητα μιας οικογένειας μπορεί να μην είναι πάντα προς το συμφέρον όλων των μελών της οικογένειας. Εάν απελάσετε κάποιος, κατά πάσα πιθανότητα απελάσετε γιατί έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα. Αν για παράδειγμα ο πατέρας είναι καταδικασμένος ε, και απελαθεί, ίσως δεν είναι προς το συμφέρον των παιδιών και της συζύγου του να απολαθούν μαζί του. Εάν η οικογένεια έχει δημιουργήσει τη ζωή της σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος, δεν θα πρέπει να τιμωρηθεί και η οικογένεια για το δικό του αδίκημα και να ε, μεταφερθούν, να πελαθούν και αυτοί μαζί του. Θα παρουσιάσω σχετική τροπολογία και ελπίζω να την υποστηρίξετε. Επίσης θα παρουσιάσω μια τροπολογία για την ε, ε, εκμάθηση γλωσσών. Θεωρώ ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι απαραίτητο τμήμα της ένταξης ε, κάποιου σε μια χώρα. Και αν κάποιος διαμένει σε μια χώρα για πέντε χρόνια, νομίζω ότι είναι λογικό να περιμένουμε να έχει μια κάποια γνώση της επίσημης γλώσσας της χώρας στην οποία διαμένει. Βέβαια θα πρέπει να εξετάσουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι βρίσκονται σε τη θέση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να προσφέρουν μαθήματα εκμάθησης και γλωσσών, καθώς επίσης και κάποια ε, επιμόρφωση ως προς τις βασικές αρχές ε, που ισχύουν σε μια χώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει ο καθένας στην κοινωνία. Για άλλη μια φορά Συγχαρητήρια και να πω ότι η ομάδα των φιλελευθέρων θα υποστηρίξει τις προτάσεις του κυρίου Μωράης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σχόλια υπάρχουν. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Congratulations, Mr. Moraes. I think... Συγχαρητήρια λοιπόν, κύριε Μωράες. Καταλάβαμε πώς έχουν τα πράγματα για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, αφού ακούσαμε και τη Βελγική Προεδρία για το τι γίνεται με το φάκελο αυτό, αλλά και με το τι γίνεται με τα υπόλοιπα συστατικά του Δουβλίνου. Τώρα, σας δίνω και πάλι το λόγο για να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, προθεσμία για τις τροπολογίες αύριο. Τετάρτη, 29 στις 12 το μεσημέρι. Κύριε Μωράης. Ναι, Πρόεδρε. Δράτω με τη ευκαιρία να πω στην ε, Προεδρία ότι μια που ο φαγγέλο αυτός είναι λίγο εκτός του πακέτου για το άσυλο, ε, εκτιμώ ότι μα έδωσαν αυτή την ενημέρωση γιατί πολλοί συνάδελφοι από όλε τι πολιτικέ ομάδε έχουν επενδύσει στο να υπάρξει πρόοδο στο πακέτο για το άσυλο. Η Προεδρία είπε ότι θα το προωθήσει από την αρχή που ανέλαβε τα καθήκοντά τη και βεβαίω και η δική μου πολιτική ομάδα θα σα ενθάρρυνε να το πράξετε. Ξέρω ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποια ερωτήματα και από άλλου εισηγητέ που εμπλέκονται στο όλο πακέτο. Σα ευχαριστώ όμω που λάβατε, κάνατε τον κόπο να μα ενημερώσετε. Ευχαριστώ και του συναδέλφου για τα πολύ κατανοητά του σχόλια, κατάλαβαν τι ήθελα να πω και έχουμε και αρκετά αισιόδοξο χρονοδιάγραμμα. Τώρα, οι τροπολογίες έχουν ως προθεσμία αύριο το μεσημέρι. Και για να σχολιάσω αυτό που είπε και η κυρία Σαρτζεντίνη, παρόλο που τώρα κουβεντιάζει με το διπλανό της, να πω ότι η κοινωτική νομοθεσία καλύπτει λέω ότι η κοινωτική νομοθεσία ε, κατά πάσα πιθανότητα καλύπτει το θέμα του απελαθέντος πρόσφυγα του οποίου η οικογένεια δεν θέλει να τον ακολουθήσει. Ας πούμε, μπορεί να υπάρξει ένα θέμα βίας ενδοοικογενειακής, μια τέτοια περίπτωση. Θα μπορούσαμε να το λύσουμε σχετικά εύκολα αυτό. Και οι υπόλοιποι συνάδελφοι έκαναν πολύ επικοδομητικές προτάσεις θα δω τι ζητούν και οι υπόλοιπε πολιτικέ ομάδε και φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία. Ε, βλέπω και στρέφομαι και προ την γραμματεία. Ε, νομίζω ότι το χρονοδιάγραμμα ε, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι σχετικά αυστηρό. Θέλουμε να ολοκληρώσουμε το θέμα αυτό μέχρι τα Χριστούγεννα. Okay. I think the is set. Ωραία. Οπότε κλείνουμε τη συζήτηση εδώ. Έχουμε την προθεσμία για τις τροπολογίες αύριο το μεσημέρι στις 12. Δεν ξέρω αν θέλει η Προεδρία κάτι να προσθέσει. Όχι. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Μωράες. Πάμε. Στο σημείο 16. για τον κανονισμό, για τον κατάλογο τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκειται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών και του καταλόγου τρίτων χωρών, οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από αυτή την υποχρέωση. Θα συζητήσουμε το φάκελο που έχει να κάνει με την απελευθέρωση της βίζας για τις θεωρήσεων για την Ταϊβάν. Λοιπόν, να δώσουμε πρώτα το λόγο στην Κομισιόν να μας παρουσιάσει την πρόταση της 5ης Ιουλίου του τρέχοντος. Μετά θα ακούσουμε το Συμβούλιο να μας παρουσιάσει τη θέση του και, αν συμφωνείτε, θα δώσουμε το λόγο και στον εισηγητή, τον κύριο Διάθ Μέρα. Και μετά βεβαίως όποιος θέλει να πάρει το λόγο Ευχαρίστω να τον ακούσουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πρώτα την Κομισιόν να μας παρουσιάσει την ε, πρόταση. Ο κύριος Γιάν Ντεκάστερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρωί σήμερα ψηφίσατε μια τροπολογία που προτείνει η Κομισιόν για τον κανονισμό 539 του 2001 που αφορά την μεταφορά της ε, Βοσνίας Ερκοβίνης και της ε, Αλβανίας από τον αρνητικό κατάλογο στο θετικό κατάλογο, από τον κατάλογο των ε, υποκείμενων σε θεώρηση χωρών στους, στον κατάλογο των χωρών που δεν υπόκειται σε αυτή την υποχρέωση. Θα θυμάστε ότι πέρσι υπήρξε άλλη μία πρόταση της Κομισιόν, συγκεκριμένα για ακόμη τρεις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, Εκεί ως Κομισιόν ακολουθήσαμε ένα πολύ συγκεκριμένο δρόμο στα πλαίσια της γενικότερου, του γενικότερου διαλόγου με τα Δυτικά Βαλκάνια για την απελευθέρωση των ε, θεωρήσεων. Η πρόταση που έχετε σήμερα θα πρέπει να ε, τη δείτε στα πλαίσια της ενδιάμεσης αναθεώρησης ε, του ε, παραρτήματος που επισυνάπτεται στον 539 του 2001. Ξέρετε ότι υπάρχουν ε, κάποια κριτήρια τα οποία πρέπει να, που, τα οποία, σύμφωνα με τα οποία ορίζονται οι ε, θετική και αρνητικοί κατάλογοι, κίνδυνοι για την ασφάλεια, κίνδυνοι για λαθρομετανάστευση, κίνδυνοι για τα εξωτερικά σύνορα της, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις εν λόγω χώρες, αμοιβαιότητα και περιφερειακή συνοχή. Πρέπει λοιπόν να ε, αξιολογηθεί το κατά πόσο οι δύο κατάλογοι αυτοί εξακολουθούν να πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Στην πρόταση Υπάρχει μια χώρα που προτείνεται να μεταφερθεί από τον αρνητικό κατάλογο στο θετικό. Οπότε να υπάρξει άρση της υποχρέωσης θεώρησης. Η Ταϊβάν είναι αυτή. Είναι πολιτική η απόφαση αυτή. Υπάρχει κι άλλο ένα θέμα, το οποίο είναι λίγο τεχνική διόρθωση ουσιαστικά στην πρόταση της Κομισιόν, για τα ε, για τις ε, νήσους, ε, για βόρειες νήσους Μαριάννα. Είναι τμήμα της, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κάτοικοι του, οι πολίτε του είναι πολίτε Ηνωμένων Πολιτειών. Οπότε και αυτοί μπορούν να εμπέσουν στην ε, άρση τη ε, θεώρηση. Οπότε θα θέλαμε οι νήσοι αυτοί να φύγουν από τον αρνητικό κατάλογο, μια που δεν είναι ξεχωριστό κράτο, οι πολίτε του είναι Αμερικανοί υπήκοοι. Τώρα, για την Ταϊβάν. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η Ταϊβάν δεν θέτει οποιοδήποτε πρόβλημα σε ό,τι αφορά την λάθρο μετανάστευση ή ε, την ασφάλεια. Τώρα, για τις εξωτερικές σχέσεις και τα σχετικά κριτήρια, πάλι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι οι γενικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ της Κίνας και της Ταϊβάν έχουν προχωρήσει πολύ, έχουν ε, αμβληνθεί εντάσεις του παρελθόντος και αυτό ήταν το κριτήριο για το οποίο η Ταϊβάν στην αρχή ήταν στον αρνητικό μας κατάλογο. Επίσης υπάρχει και το θέμα της περιφερειακής συνοχής. Ήδη κάποιες χώρες της περιοχής όπως η Νότια Κορέα, η Ιαπωνία ε, δεν υπόκεινται στην ε, υποχρέωση θεώρησης οπότε αυτή η πρόοδος θα, θα προσφέρει στην περιφερειακή συνοχή. Τελευταίο ε, κριτήριο αμοιβαιότητα. Προς το παρόν η Ταϊβάν εξακολουθεί να θέτει υποχρέωση θεώρησης για τρία κρατημέλη μας, Κύπρο, Ρουμανία, Βουλγαρία, αλλά έχει δεσμευθεί να άρει τις, υποχρέωσεις, τις απαιτήσεις θεώρησης για αυτά τα τρία κρατημέλη. Και δεσμεύτηκε επίσης να αυξήσει την, ε, την διαμονή από 30 μέρες σε 90 μέρες. Σήμερα η, θεώρηση ε, επιτρέπει την ε, παραμονή για 30 μέρες. Θα ζητήσουμε λοιπόν από τους ε, Ταϊβανέζους ομολόγους μας να επιβεβαιώσουν σε αυτή τους τη δέσμευση, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πλήρης αμοιβαιότητα. Αυτά, Πρόεδρε, ε, εν συντομία, στην, στο Συμβούλιο έχει ξεκινήσει η δουλειά επί της πρότασης αυτής. Ε, Μπορεί να υπάρχει ένα θέμα για το οποίο ίσως να υπάρξει μια τροπολογία, αλλά θα το αφήσω στην Προεδρία να σας το εξηγήσει περί τίνος πρόκειται δηλαδή. Και βεβαίως μετά, εάν θέλετε, μπορώ να σχολιάσω αν προταθεί κάποια τροπολογία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρουσίαση της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τώρα να ακούσουμε τη Βελγική Προεδρία. Η Βελγική Προεδρία θέλει το λόγο. Ο κύριος Εμίλ, η, κυρία, συγγνώμη, διορθώνει ο πρόεδρος, η κυρία Εμίλ Μπρέιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Όπως ε, θα έχετε ήδη ακούσει, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τμήμα τη συνήθους αναθεώρησης του κανονισμού 539 του 2001. Πέραν των κριτηρίων που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να προσθέσω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας πούν ποιες χώρες θεωρούν ότι είναι έτοιμες να μπουν στο θετικό κατάλογο και, δεν, ε, ε, και αντίστοιχα ποιες χώρες ε, δεν πληρούν τα κριτήρια και θα πρέπει να μπουν στον αρνητικό κατάλογο. Το θέμα των κρατών μελών είναι σημαντικό και οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν επεπισμένες ότι η Ταϊβάν έπρεπε να μπει στον κατάλογο, γι' αυτό και εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. η Κομισιόν θέλει να τροποποιήσει την πρόταση για την Ταϊβάν Άνω των 60.000 Ταϊβανέζων δεν ζουν στην Ταϊβάν, αλλά ζουν στο εξωτερικό και εκεί ε, ε, για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχουν διαφορετικά διαβατήρια από τους, ε, σε σχέση με τους κατοίκους που διαμένουν στην Ταϊβάν μόνιμα. Τα διαβατήρια αυτά δεν τους επιτρέπουν να μεταβούν στην Ταϊβάν χωρίς θεώρηση. Για κάθε λοιπόν ταξίδι τους ε, στην Ταϊβάν πρέπει να λάβουν πρώτερη έγκριση από τις ε, αρχές της Ταϊβάν. Δεν θεωρούμε λογικό να δίνουμε θεωρήσεις και διευκολύνσεις θεώρησης σε αυτή τη συγκεκριμένη κατηγορία και γι' αυτό το Συμβούλιο θα ήθελε να γίνει και μια σχετική τροποποίηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κυρίως με τον εισηγητή, με τον κύριο Διαυτεμέρα, ώστε τα θέματα διευκόλυνσης θεωρήσεων για την Ταϊβάν μπορούν να υιοθετηθούν το συντομότερο δυνατόν. Ε, ελπίζουμε πριν από το τέλος του έτους. Ευχαριστώ την κυρία Μπρέιν και τώρα να ακούσουμε τον εισηγητή, ο κύριο Διαθεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με πολύ προσοχή την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την άποψη του Συμβουλίου και σε γενικές γραμμές συμφωνώ απολύτως με τα κριτήρια που ανέφεραν. Σήμερα θα κάνω μια συνοπτική παρουσίαση της έκθεσής μου και η εκτεταμένη παρουσίαση θα γίνει στην ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας στις 11 Οκτωβρίου, κύριε Πρόεδρε. Θεωρώ ότι είναι δεδομένες οι πληροφορίες που ακούσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο και προσθέτω τα εξή. Η κατάσταση στην Ταϊβάν δεν αποτελεί καμία απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε σε θέματα νόμιμης μεταμάστευσης, ούτε σε θέματα δημόσιας ασφάλειας. Όπως ε, θα δείτε από τις ενδελεχέστατες πληροφορίες που θα έχουμε στην τελική έκθεση, η ε, Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Ταϊβάν ε, έχουν βιώσει μια πολύ υψηλή οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, φτάνοντας ένα κατακεφαλήν εισόδημα άνω των 30.000 δολαρίων ετησίως και το ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2010 ήταν 5,2% πολύ κατώτερο, όπως ε, πολύ λογικά καταλαβαίνουμε, από το σύνολο των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι το ποσοστό ενεργείας είναι στο 10,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τους λόγους αυτούς ε, θεωρούμε ότι η Ταϊβάν δεν αποτελεί κίνδυνο σε θέματα παράνομης μετανάστευσης ή σε θέματα νόμιμης μετανάστευσης. Ως παράδειγμα να σας υπενθυμίσω τα στοιχεία που μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006-2008 στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε μόνο 45 παράνομους μετανάστευς από την ε, Ταϊβάν. Ταυτόχρονα η Ταϊβάν απαλλάσσει από το καθεστώς θεώρηση όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εξαίρεση τριών χωρών όπως αναφέρθηκε ήδη, την Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Αλλά για τις τρεις αυτές χώρες η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνα δεσμεύτηκε επισήμω και αυτό μου είπαν οι εκπρόσωποι των αρχών της Κίνας στις Βρυξέλλες να εγκρίνει την πλήρη απαλλαγή θεώρησης για τις τρεις χώρες αυτές πριν από το τέλος του έτους. Επίσης, συμφωνώ με αυτό που ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι θα πρέπει να ζητήσουμε και να λάβουμε αυτή τη δέσμευση γραπτός. Πρόκειται για μια κατάσταση την οποία θα ήθελα να γνωρίζετε. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έκαναν απαλλαγή των θεωρήσεων για την Κίνα το Μάρτιο και τον Ιούλιο του 2009 αντίστοιχα. Για άλλες χώρες, για την ε, ε, Νότια Κορέα, τη Σιγκαπούρη, τη Νέα Ζηλανδία, είχαμε και πάλι απαλλαγή από τη θεώρηση ε. και για τον τομέα της ασφάλειας θα πρέπει να πούμε ότι τα ταξιδιωτικά έγγραφα της Ταϊβάν και αυτό το διαπίστωσα η διεισόμαση καλύπτουν όλες τις προδιαγραφές που απαιτούν ο, η ΙΑΤΑ και περιλαμβάνουν και κάποια επιπλέον στοιχεία τα οποία είναι πολύ προηγμένα για την καταπολέμηση της παραποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει απαλλάξει από τις θεωρήσεις άλλες χώρες ε, της περιοχής, ε, το Χονγκ Κόνγκ, το Μακάο, την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη. Ως προς την εφαρμογή της αρχής της εδαφικής συνοχής και της, ε, των πολιτικών υποστήριξης από κοινοτικής πλευράς, θα πρέπει να είμαστε υπέρ της επίτευξης του στόχου αυτής της πρότασης, όπως μόλις σας είπα. Σε γενικές γραμμές, η συμπερίληψη της Ταϊβάν στο θετικό κατάλογο θεωρείται ότι είναι η πλέον δεδειγμένη λύση και μάλιστα απαραίτητη. Επίσης, αναφερθήκαμε και Στα νησιά Μαριάνας του Βορρά οι πολίτες αυτοί είναι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως ε, δεν θα πρέπει να βρίσκονται στο παράρτημα 1 του κανονισμού. Και επίσης θα, δεν θα πρέπει να πετούμε από αυτούς τους πολίτες ε, να λαμβάνουν θεώρηση για να ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εξέτασε το θέμα αυτό και έχει ήδη δώσει θετική γνώμη. Όσον αφορά τώρα την τροποποίηση που θα παρουσιάσουν οι χώρες μέλη στην πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπή με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Έχω ενδελαχέστατε πληροφορίες για το διαβατήριο της διασποράς και στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ταϊβανέζικο διαβατήριο για τους Κινέζους που βρίσκονται ε, πέραν της Ταϊβάν. Δεν είναι εγγεγραμμένη στα Μητρώα της Ταϊβάν και η, διάκριση αυτή αφορά περίπου 65.000 Ταϊβανέζους. Έχω εδώ μπροστά μου την τροποποίηση που προτείνει το Συμβούλιο που λέει ότι η εξαίρεση της ε, υποχρέωσης θεώρησης δεν αφορά τους πολίτες ε, που έχουν διαβατήρια τα οποία ε, έχουν εκδοθεί από τις αρχές του Ταϊβάν και, της Ταϊβάν και δεν περιλαμβάνουν και αριθμό ταυτότητας. Συνήθ, ε, πρόκειται για περίπου 65.000 ανθρώπους. Εγώ τη δέχομαι αυτή την ε, τροποποίηση και θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι οι κινέζικες αρχές ε, δεν έχουν πρόβλημα με αυτή την τροποποίηση, δεν θα ζητήσουν κάτι ως αντάλλαγμα. Και ε, νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι με αυτό μπορώ να ολοκληρώσω την ε, παρουσίασή μου και θα ήθελα να ζητήσω πριν κλείσω τα εξή. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών νομίζω ότι μπορεί να ξεκινήσει από σήμερα. Αναφερόμαστε στην ε, πρόταση τροποποίηση του κανονισμού και θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 12 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα μετά από την επίσημη παρουσίαση της έκθεσής μου Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να ζητήσω από όλη την Επιτροπή να υποστηρίξει την πρότασή μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διαθεμέρα. Ο κύριος Μπρόντς θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Να πω ότι οι πολίτες τρίτων χωρών δεν χρειάζονται πλέον θεώρηση. Αυτό συνήθως λένε ότι βοηθά κόσμο και ότι είναι ή φοιτητέ ή τρομοκράτε. Αλλά ίσω να μην είναι ο κατάλληλο τρόπο να του εμποδίσουμε να δουλέψουν ή να φτιάξουν το σπιτικό του. Ο εισηγητή μίλησε για τον ελάχιστο νούμερο αριθμό Ταϊβανών που ε, είναι εδώ και δουλεύουν ω ως ε, μετανάστε, αλλά δεν έδωσε αντίστοιχα νούμερα για καμιά άλλη χώρα. Ούτε στην ε, λευκή λίστα, ούτε στη μαύρη λίστα. Τώρα, μια έλλειψη μιας άδεια εργασίας μπορεί να τους ε, ε, εμποδίσει να μπουν στην επίσημη αγορά, αλλά δεν τους εμποδίζει αυτό καθόλου από το να μπουν στην ανεπίσημη αγορά, που δεν ισχύει κανένας νόμος. Και τέτοια οι άνθρωποι μπορεί να πέσουν θύματα της χειρότερης εκμετάλλευσης. Επιπλέον, ε, έρεται η ανάγκη για θεώρηση για τις χώρες ε, που υπέγραψαν την Συμφωνία Σέγγεν. Αλλά αυτό συμπεριλαμβάνει και την, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, ε, ξεπερνούν, ξεπερνάει η ευφυΐα και η πανουργία των ανθρώπων, τους, τα εμπόδια και τους περιορισμούς για να έρθουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστώ, κύριε, ο κύριος Μπουσούτιλ. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε για να πω στο τελευταίο μιλητή, αν κατάλαβα καλά, το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχει απελευθερώσει την ρίζα για την Ταϊβάν, άρα απλώ ακολουθούμε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν ισχύει το αντίστροφο. τώρα, εγώ θέλω να παρέμβω για να στηρίξω αυτή την πρόταση. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να αρθεί η χορήγηση βίζας στην Ταϊβάν για διάφορους λόγους. Η Ταϊβάν είναι ευημερή χώρα. Έχει οικονομική ανάπτυξη τρομερή, πάνω από 10% φέτος. Ε, είναι στο προς και του τουριστικού τομέα μας βέβαια το να άρουμε την υποχρέωση βίζας διότι θα αυξηθούν οι τουρίστες από αυτή τη χώρα. Αυτό ήδη ε, συνέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήρε την υποχρέωση βίζας και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη ως Ευρωπαίοι πολίτες δεν απαιτούμε θεώρηση Μάλλον δεν χρειάζεται θεώρηση για μα για να πάμε στην Ταϊβάν. Βέβαια υπάρχει εξαίρεση τη Κύπρου, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όπω ακούσαμε και με χαρά ακούω ότι και αυτές οι χώρες δεν θα χρειάζονται σε λίγο βίζα. Υποστηρίζω λοιπόν τον εισηγητή και ελπίζω να γίνει όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ κύριε Μπουσούτιλ. Άλλα σχόλια. Θέλει κάποιο να σχολιάσει. Ναι. Ναι, γνωρίζω ότι, γιατί ακούσαμε από την Κομισιόν ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ήδη έχει άρει την υποχρέωση βίζας για την Ταϊβάν. Τα σχόλιά μου δεν αφορούσαν μόνο την Ταϊβάν, γιατί ο εισηγητή ε, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα παράνομη μετανάστευση. Εγώ είπα γενικότερα για τι χώρε που είναι στον θετικό κατάλογο. Now. There Άλλα σχόλια. Δεν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο. Κύριε Ντίας Δεμάρα, κύριε Σιγητά, θέλετε να κάνετε κάποια σχόλια. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, κυρίως τον κύριο Μπουσουτήλ και για την παρέμβαση του κυρίου Μπρόνς. Δεν έχω τίποτα να πω διότι στη δεύτερη παρέμβασή του ούτως ή άλλως διευκρίνησε ότι δεν αναφερόταν απλώς και μόνο στην Ταϊβάν. Αυτό που σκόπευα να πω, αλλά δεν θα το πω, θα το πω την επόμενη φορά που θα μιλήσω, είναι να αναφερθώ εκτεταμένα στους οικονομικούς δείκτες της Ταϊβάν που είναι από τους καλύτερους στον κόσμο και να πω ότι από την πείρα που έχουμε οι Ταϊβανέζοι έρχονται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο πολύ για τουρισμό και για να αφήσουν συνάλλαγμα παρά για άλλους λόγους όπως πιστεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία για να εργαστούν. Νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό και για τις δύο πλευρές να τους απαλλάξουμε από τις θεωρήσεις ε, για το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τίεστε Μέρα. Μπορούμε λοιπόν, με βάση τα όσα μας είπε και ο εισηγητής, ο κύριος Μέρα, να συζητήσουμε τις προθεσμίες. Κατάθεση τροπολογιών Αμέσως μετά την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στις αρχές Οκτωβρίου θα παρουσιάσουμε την έκθεση στι 11 Οκτωβρίου στη συνεδρία τη Επιτροπής, προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 12 Οκτωβρίου το μεσημέρι. be opening way for a vote late October. Θα ψηφίσουμε λοιπόν κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη Οκτωβρίου στη συνεδρία της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και στη συνέχεια στην Ολομέλεια του Νοεμβρίου θα μπορούσαμε κάλλιστα να ψηφίσουμε στην ε, Ολομέλεια. Αν συμφωνείτε, αυτό θα κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, έχουμε ένα ακόμα σημείο, το υπαριθμό 17, πριν ολοκληρώσουμε τη σημερινή συνεδρίαση ο Οργανισμός για τη Λειτουργική Διαχείριση Μεγάλων Πληροφοριακών Συστημάτων στον τομέα της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εισηγητής ο κύριος Κοέγιο. Έχουμε λίγα λεπτά στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε τις τροπολογίες που κατατέθησαν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ ε, για το σχέδιο έκθεσης του κυρίου Κοέλιο για τον οργανισμό της λειτουργικής διαχείρισης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων. Θα ακούσουμε λοιπόν πρώτα τον κύριο Κοέλιο, μετά τους λοιπούς συναδέλφους που θέλουν να λάβουν το λόγο για τη συζήτηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη Βελγική Προεδρία. Καταρχάς, In our next meeting... να σας πω ότι στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία είναι για τις 11 Οκτωβρίου έχουμε ψήφο προσανατολισμού για το θέμα αυτό. Κύριε Κοέλιο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα όπως πάντα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Να ευχαριστήσω για τη συνεργασία σας και για το γεγονός ότι με τις προτάσεις σας εμπλουτίσατε την έκθεσή μου. Εγώ συνεδρίασα μαζί τους ε, χτες και καθορίσαμε, κα, κα, καταλήξαμε μάλλον σε κάποιες συμβαστικές ε, τροπολογίες που θα σταλούν σε όλους τους συναδέλφους και που, όπως θύμισε και ο Πρόεδρος, τις επόμενες μέρες, 11 Οκτωβρίου δηλαδή, θα τις ψηφίσουμε. Οι συμβαστικές τροπολογίες βασικά αφορούν που ήδη έχουμε συζητήσει εδώ επανελειμμένως και είναι ανησυχίες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και του Ευρωκοινοβουλίου. Και κυρίως στόχο έχουμε να αποφύγουμε μέσω πιλωτικών προγραμμάτων να αλλάξουν οι στόχοι του οργανισμού χωρίς την, τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπογραμμίσουμε ποιες είναι οι αποστολές του οργανισμού και να εγγυηθούμε ότι αυτές εντάσσονται στους στόχους μας. και να δοθεί μια ιδιαίτερη ε, προσοχή στην προστασία των δεδομένων. Επιπλέον ένα σύνολο προϋποθέσεων για την επιλογή της τοποθεσίας του οργανισμού. Όπως είπα στην αρχή, δεν έχουμε την νομική άποψη ότι αυτό είναι θέμα του Συμβουλίου, αλλά ότι το Κοινοβούλιο δεν επιθυμεί να αποτελέσει έναν πόλο προβλημάτων. Δεχόμαστε το τι θα πει το Συμβούλιο από τη στιγμή που αυτό σέβεται ένα σύνολο προϋποθέσεων που απαριθμούνται στο εγγραφό μας. Αυτά, Πρόεδρε, είμαι στην διάθεση των συναδέλφων αν θέλουν να θέσουν ερωτήσεις για τις ε, προτάσεις, τις συμβαστικές μας. Εξάλλου πρόκειται για διάφορα θέματα τα οποία ήδη έχουμε συζητήσει επανελειμμένως στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ κύριε Κουαΐου. Τώρα θα ακούσουμε την Βελγική Προεδρία. Ευχαριστώ, κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει συζήτηση αυτή και σε επίπεδο ομάδα υπάρχουν βεβαίω ακόμη κάποια εκκρεμή θέματα, αλλά θεωρούμε ότι η περαιτέρω συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών θα μας ε, δώσει τη δυνατότητα να συντονίσουμε καλύτερα τη δουλειά μας, γιατί μας ενδιαφέρει φυσικά πάρα πολύ να δούμε ποιες θα είναι οι τροπολογίες. Και βεβαίως ε, εάν ε, υπάρξει και ψηφοφορία, ελπίζω να καταφέρουμε να καταλήξουμε και σε μια ε, λύση που να ικανοποιεί όλους. Ευχαριστώ κύριε Βαμπέλα. Τώρα περνούμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Τουντουράχε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ο εισηγητής είπε ότι ήδη το έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό αρκετές φορές και στην Επιτροπή εδώ και την ουσία της πρότασης και τις περισσότερες εκ των τροπολογιών. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε και η Προεδρία, θα συμφωνήσω και με αυτά που είπε στην εισαγωγή του εισηγητής. Έχει γίνει πραγματικά εξαιρετική πρόοδος. Οι περισσότερες από τις τροπολογίες θα βελτιώσουν το κείμενο και τις καλωσορίζουμε δεν θα σχολιάσω τα όσα είπαμε σε παλαιότερες συνεδριάσεις, απλώς θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για τις νέες τροπολογίε που έχουν υποβληθεί πρόσφατα το πιλωτικό πρόγραμμα ήταν κομμάτι μια ε, συγκεκριμένη τροπολογία που την ανέφερε ο εισηγητή. Ο τρόπο με τον οποίο το έχει συντάξει η Κομισιόν, μάλλον που έχει καταλάβει η Κομισιόν το κείμενο, δεν θεωρούσαμε ότι ε, θα προσθεθούν οι στόχοι ή τα πιλωτικά προγράμματα αυτά στου ε, στόχου ή ότι θα αποτρέψουν τον οργανισμό από το να κάνει οτιδήποτε. Απλώ τα πιλωτικά προγράμματα είναι απαραίτητα, είναι εργαλεία εφαρμογή του προπολογισμού, τα οποία χρησιμοποιεί πάντα η Κομισιόν όταν χαράσει πολιτική και νομοθεσία. Ε, αυτό είναι ούτως ή άλλως κάτι που βασίζεται και στο άρθρο 49 του οικονομικού α, κανονισμού. Οπότε δεν είναι κάτι καινούριο που θα χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση αυτή του οργανισμού ούτε για να ε, προσθέσει κάτι, ούτε για να εφαρμόσει οποιαδήποτε νέα προγράμματα. Είναι τμήμα, σας λέω και πάλι, της όλης προετοιμασίας της πολιτικής και της νομοθεσίας που οραματίζεται η Κομισιόν σε αυτόν τον νέο τομέα και όχι ένα ξεχωριστό πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο βεβαίω παραμένει στη διακριτική ευκαιρία τη Κομισιόν να εκπονήσει. Αλλά παρόλα αυτά ε, η Κομισιόν έχει μεγάλη προγνωμοσύνη στον τομέα αυτό και θεωρήσαμε ότι αυτά τα προγράμματα είναι αξιόπιστα για να τα χρησιμοποιήσει και ο οργανισμό. Βεβαίω στα πλαίσια και τη διαφάνεια δεχτήκαμε τι προτάσει που έγιναν ε, σε σχέση με τι πρώτε πληροφορίε που είχαμε για τα πιλωτικά αυτά προγράμματα και από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική άποψη όλων των ενδιαφερομένων ε, φορέων. Παρ' όλα αυτά, ε, τα πιλωτικά αυτά προγράμματα ε, βασι... δεν θέλαμε να, είναι, ε, να εξαρτώνται απόλυτα από τις αποφάσεις ε, τη, του, ενός του άλλου θεσμικού οργάνου γιατί έτσι υπονομεύεται η δική μας λειτουργία όταν αφορά την εφαρμογή του οικονομικού κανονισμού και του προπολογισμού. Έγινε λοιπόν ε, αρκετή προετοιμασία κατά τη διάρκεια της υποβολής της πρότασης. Ε, υποστηρίζουμε φυσικά αυτές τις ε, απαιτήσει και μια που το είπε και ο εισηγητής, θεωρώ ότι αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση που πρέπει να την πάρει το Συμβούλιο. Τώρα να προσθέσουμε νέες απαιτήσει πριν από την έγκριση του κειμένου ξέροντας ότι η απόφαση για τον, για τον οργανισμό θα πρέπει επίσης να ληφθεί πριν από την υιοθέτηση του κειμένου δεν νομίζω ότι θα είναι ιδιαίτερο αποτελεσματικό για την ίδια την απόφαση. Υπάρχει η τροπολογία 65 για την εισαγωγή της, του διαχωρισμού μεταξύ του πλάνου ασφάλειας και του πλάνου ενημέρω, ενημέρωσης και ασφάλειας. Ε, όλα αυτά είναι κομμάτι της ίδιας ιδέας η ασφάλεια των ε, προγραμμάτων πληροφορική. Είτε είναι φυσική η ασφάλεια του, του ε, κτηρίου μέσα στο οποίο βρίσκονται, είτε είναι η ασφάλεια των πληροφοριών που επεξεργάζονται αυτά τα συστήματα. Όλα αποτελούν τμήματα μιας, ενός σχεδίου που θα πρέπει να υιοθετήσει ο οργανισμός. Οπότε, εμείς δεν θα θέλαμε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των δύο αυτών ε, όρων, γιατί είναι τμήματα του ιδίου οράματος. οράματος. Τώρα, για το ΕΝΙΣΑ και την ε, συμπερίληψή του στην, ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην, ε, στα πιο ουσιαστικά, στην πιο ουσιαστική λειτουργία το, του οργανισμού. Φυσικά γνωρίζουμε την εντολή που έχει ο ΕΝΙΣΑ. Είναι ένας οργανισμός που είναι συμβουλευτικός για την ασφάλεια των δικτύων και θα θέλαμε να υπάρχει μία διάταξη που να ενισχύει τη δυνατότητα που έχει ο διευθυντής να διαβουλεύεται, να συμβουλεύεται όποιον θεωρεί κατάλληλο. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε την εντολή που έχει ο ΕΝΙΣΑ και ούτε βέβαια και το πεδίο μέσα στο οποίο δρά και συμβουλεύει ε, ο οργανισμός αυτός. Τώρα, η συχνότητα των αξιολογήσεων. Ε, με τις τροπολογίες έχει πάει στα τρία χρόνια. Θεωρούμε ότι είναι πολύ μικρό το χρονικό αυτό διάστημα. Καταρχήν δεν υπάρχει προηγούμενο. Ε, το, για, τις, για τους υπόλοιπους οργανισμούς ισχύουν τα πέντε χρόνια. Και πέρα από αυτό υπάρχει και το θέμα του πεδίου εφαρμογής αυτών των αξιολογήσεων. Ε, υπάρχουν και κάποιε τροπολογίε που αφορούν την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να επαφείται στο EDPS ε, και στι αρμοδιότητές του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρξει κάποια υπεργολαβία εδώ από κάποιον που θα κάνει αυτή την αξιολόγηση γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξει επικάλυψη αρμοδιοτήτων μεταξύ του EDPS και του εξωτερικού συνεργάτη που θα αναλάβει να κάνει τι ε, αξιολογήσει. Αυτά, Πρόεδρος, απάντηση για τις νέε τροπολογίε. Φυσικά Κατανοώ ότι υπάρχουν και κάποιε ε, αναθεωρημένες τροπολογίε, Θα ήθελα να τι δω και βεβαίω να απαντήσω και σε μεταγενέστερες συζητήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλβαρο. Thank you Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Άκουσα τα όσα είπε η Κομισιόν και το Συμβουλίο, ο Καρλός Κοέγιος στην καθοδήγησε πολύ συνετά του συντονιστέ σε αυτό το φάκελο και θεωρώ ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε που υπέβαλε χτε δεν θα έπρεπε να αποτελέσουν κανένα πρόβλημα για να ψηφιστεί η έκθεσή του. Τα θέματα που θίγει φυσικά τα συμμεριζόμαστε ω πολιτική ομάδα. Ε, ενδιαφέρον όμω θα ήταν να δούμε και τα θέματα που ανέφερε η Κομισιόν και τα οποία εμπλέκουν και τον ΕΝΙΣΑ και άλλα θέματα, γιατί ούτως ή άλλως είναι θέματα τα οποία, από τα οποία περιμένουμε περαιτέρω εξελίξεις. Επίσης, θα ήθελα να ακούσω από την Κομισιόν ή από το Συμβούλιο το εξή. Μου είπανε ότι, επειδή είμαι και μέλο τη Επιτροπή Προπολογισμού, ότι στον προπολογισμό για, τα, για του μεγάλου οργανισμού πληροφορική υπάρχει ένα ποσό αποθεματικό για την μετάπτωση του ε, συστηματος συς SIS-2 για να ενταχθεί στο, στη λειτουργία του οργανισμού αυτού. Ισχύει αυτό γιατί στην αρχική πρόταση δεν το βρίσκουμε αυτό πουθενά. Και δεύτερον, για, σχετικά με το τι γίνεται τώρα με το ΣΥΣΔΙΟ, 2 θα, θα, ξανα, θα προχωρήσει αυτό, θα είναι λειτουργικό, ακόμη και αν δεν ολοκληρωθεί το ΣΥΣ 2 θα προχωρήσει το υπόλοιπο σύστημα. Ε, εν πάση περιπτώσει θα είναι ίσως, αν δεν γίνουν όλα αυτά, ίσως αυτό που λέει ο Κάρλος να είναι περιττό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Κάρλος Κοέλιο για την δουλειά του και τους άλλους κοιόδες. Ήταν πολύ καλή δουλειά, έχουμε καλό αποτέλεσμα. Να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις για να τις ακούσει και το η Κομισιόν και το Συμβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό νομίζω ε, τα όσα εμείς αναφέρουμε ως ανησυχίες και ως επιχειρήματα για όλη αυτή την υπόθεση του οργανισμού για το πώς τα συστήματα αυτά συνδυάζονται από τεχνικής άποψης και πιστεύω πως αυτό είναι και πάρα πολύ σημαντικό να, να ισχύσει και για τις μελλοντικές συζητήσεις δηλαδή Δηλαδή ότι ανησυχούμε ιδιαίτερα όσον αφορά τις τάσεις που υπάρχουν για διαλειτουργικότητα μεταξύ των βάσεων δεδομένων. Νομίζω πως ε, πάντα θα πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις από το Κοινοβούλιο όταν αλλάζει κάτι σε αυτές τις υποδομές. Πολύ ισχυρό μήνυμα από το Κοινοβούλιο λοιπόν θα πρέπει να δοθεί και θα πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους που ενέχουν οι κεντρικές βάσεις δεδομένων και τα συστήματα πολύ μεγάλης κλίμακας. Εγώ πάντοτε διστάζω όσον αφορά την, κέντρο, και την συγκέντρωση υπερβολικά πολλών στοιχείων, γιατί ο κίνδυνος είναι ο μεγαλύτερος. Αυτή είναι μια γενική παρατήρηση που πρέπει πάντοτε να λαμβάνετε υπόψη όταν δουλεύουμε με αυτό το σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη δουλειά αυτή. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Κυρία Γκυγιόμ, εγώ θα είμαι ακόμη πιο σύντομη να επενέσω κι εγώ τον ε, Κουέλιο για τον τρόπο με τον οποίο μας κάλεσε και μας έτεινε το χείρα συνεργασίας. Τώρα για το θέμα ε, της αρμοδιότητας ε, της υπηρεσίας, ε, στόχος δεν είναι η διαλειτουργικότητα των δεδομένων, ούτε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής, αυτό θα είναι από ad hoc απόφασης, ή ακόμα κάποιες απαιτήσεις όσον αφορά την έδρα, δηλαδή ζητήματα τα οποία είχαμε θίξει στην ομάδα μας και υπό τη μορφή τροπολογιών, και ε, θέματα τα οποία βρίσκουμε μέσα στις συμβαστικές τροπολογίες που είδαμε και εξετάσαμε εχθές. Νομίζω λοιπόν πως μπορούμε να είμαστε θετικοί για αυτό την έκθεση. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Έρμστ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολλά ακούστηκαν ε, ήδη για τα προβλήματα που υπάρχουν. Ε, θα ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Κοέλιο. Κατάφερε να συνθέσει πολλές ε, διαφορετικές προτάσεις, τροπολογίες. Πραγματικά είναι πολύ αξιόλογη η πρότασή του. Θα ήθελα δύο πραγματάκια όμω να πω για να τα σκεφτούμε. Καταρχήν, αν δούμε την γνωμοδότηση τη Επιτροπή Προπολογισμού, υπάρχουν πάρα πολλά εκκρεμή ερωτήματα τα οποία τελικά δεν έχουν λάβει απάντηση. Ε, ας πούμε, αναλύσεις κόστου ωφέλειας, συγκεκριμένες προοπτικές για τον προπολογισμό. Ε, δεν νομίζω ότι είναι επαρκές αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμή ως προς αυτά και νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε περισσότερο υπόψη μας. Επίσης, ο δικός χάρτης για την περαιτέρω ανάπτυξη των συστημάτων, ε, ανάλυση χρηστικότητας, θα μπορούσαμε να την κάνουμε. Ε, ήδη στην γνωμοδότηση ζητείται συνέχεια το κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό το project και κατά πόσο θα πρέπει όντω να δημιουργηθεί αυτό ο οργανισμό. Αυτό είναι ένα το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά. Δεύτερον, η συμπερίληψη περαιτέρω μεγάλων συστημάτων πληροφορικής και το ερώτημα πώς θα ρυθμίσουμε έναν τέτοιον οργανισμό αν δηλαδή δεν προκύψει, δεν καταλήξουμε στο ΣΥΣ2, τι θα γίνει σε τέτοια περίπτωση. Θα ήθελα λοιπόν να το δούμε και αυτό. Μήπω χρειαζόμαστε μια εναλλακτική λύση. Αν δεν προκύψει το ΣΥΣ2. Ε, ορισμός ο, ο περιορισμός συγγνώμη, των α, ε, ε, συστημάτων πληροφορικής νομίζω είναι, είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. και νομίζω ότι ίσως θα έπρεπε να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Ε, τα υπόλοιπα ε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να τα αναφέρω, ούτως ή άλλως έχουν συζητηθεί και σε άλλα επίπεδα. Ε, ευχαριστώ για το χρόνο σας και ευχαριστώ τον εισηγητή. Εγώ ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Ωραία. Κύριε Κοέλιο, εσείς? Thank you to uh, uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους συναδέλφους. Να τους ευχαριστήσω για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε σε αυτό το δύσκολο ντοσιέ. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα σχολεία της. Ορισμένε ε, από τι τροπολογίε έχουν ήδη αντικατασταθεί από συμβιβαστικέ, οπότε δεν χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε δυσκολίε. Για παράδειγμα, συμμετοχή άλλων θεσμών ή υπηρεσιών ή οργανισμών στην διαχείριση αυτού του οργανισμού. Έχουμε ένα πρόβλημα ωστόσο. Στην Επιτροπή Προπολογισμού ασκείται μεγάλη πίεση για περιορισμό του κόστους και του τρόπου διαχείρισης. Δεν είμαι κατά αυτής της ιδέας, αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι έχουμε να κάνουμε θέματα που σχετίζονται με την κυριαρχία και τον έλεγχο του προπολογισμού όλων των κρατών μελών. Και γι' αυτό το λόγο δεν νομίζω πως θα ήταν σοφό να περιοριστεί ο αριθμός των ε, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι να μην μπορούν όλα τα κράτη-μέλη να συμμετέχουν. Αλλά οι συμβαστικές τροπολογίες που κάναμε χτες θα σταλούν σε όλους και έτσι θα έχουν όλοι την ευκαιρία να τις δουν και να τις σχολιάσουν. Τελευταία παρατήρηση, Πρόεδρε, αφορά τα σχόλια της Κομισιόν για τους όρους. Είναι αλήθεια ότι το Συμβούλιο θα αποφασίσει για την τοποθεσία και αυτό θα μπει μέσα στο κείμενο. Ώστε να μπορούμε να πούμε οι όροι δεν χρειάζονται, αλλά Έχουμε να κάνουμε μια διαδικασία συνεργασίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Και το Συμβούλιο θα ξέρει όταν θα λάβει αυτή την απόφαση ποιοι είναι οι όροι μας. Διότι αν δεν τηρηθούν οι δικοί μας όροι, δεν θα συμφωνήσουμε να βάλουμε αυτή την τοποθεσία στο κείμενο. Προσπαθούμε με καλή διάθεση να συνεργαστούμε με το Συμβούλιο, αλλά δεν πρόκειται να εγκρίνουμε οποιαδήποτε λύση. Μία λύση που θα συμφωνεί με τις δικές μας ανησυχίες, ναι. Δεν θέλουμε να είμαστε κομμάτι του γεωγραφικού πολέμου, δεν είναι δικό μας το πρόβλημα το να πάει σε μια χώρα ή μια άλλη, αλλά θέλουμε ή τοποθεσία να σέβεται τους κανόνες και τους όρους που έχουμε θεσπίσει. Και γι' αυτό και έχουμε και σχετικό άρθρο. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Coelho. If no further comments from the Commission or the Presidency, would, the Commission or the Presidency... Η Κομισιόν, η Προεδρία θέλουν να πούν κάτι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Πριν ε, απαντήσω στις ερωτήσεις των σχεδόν εισηγητών. Εγώ θέλω να στηρίξω τα όσα είπε ο κ. Κουέλιο νωρίτερα για τη σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι κάτι που έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή προπολογισμού, στη στιγμή της συζήτηση των τροπολογιών εκεί. Εμείς κατανοούμε την ανάγκη για περικοπή του κόστου, αλλά όπω είπε και ο κ. Κουέλιο, η ιδιαιτερότητα αυτού του οργανισμού είναι τέτοιο που κάθε μέλος πρέπει να έχει έναν εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί είναι τα κράτη-μέλη οι ιδιοκτήτες των στοιχείων που επεξεργάζεται το σύστημα. Άρα πρέπει να έχουν ένα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο. Τώρα, για το ερώτημα κατά πόσο χρειάζεται υπάρχει κόστος για την SIS και ένα στην sis 2 αν, υπάρχει κόστος για τη μεταφορά των στοιχείων. Όχι, δεν υπάρχει κανένα κόστος ε, το οποίο να μπαίνει μέσα στην προϋπολογισμό της υπηρεσίας του οργανισμού. Το SIS2, το SIS2 και η ε, αντίκτυπο στην οργανισμό, μια άλλη παρατήρηση ενός άλλου βουλευτή, και πάλι η απάντηση είναι όχι, δεν υπάρχει τίποτα που να επηρεάζει τον οργανισμό από το ΣΥΣ2. Δεν είναι οργανισμός του, του ΣΥΣ2, είναι ένας οργανισμός που θα πρέπει να λειτουργεί για όλα τα συστήματα που υπάρχουν στον τομέα της δικαιοσύνη, της ελευθερίας και της ασφάλειας και τα μελλοντικά συστήματα επίσης. Έχουμε και το Eurodac, το οποίο θα αναλάβει ο οργανισμός, το ΒΙΣ επίσης ε, και το ΣΥΣ σε οποιαδήποτε τεχνική μορφή μέχρι τότε θα είναι ευθύνη της Κομισιόν και όταν το ΣΥΣ 2 θα είναι έτοιμο τότε ο οργανισμός θα αναλάβει τον έλεγχο της λειτουργίας αλλά όπως είπα, ό,τι και αν γίνει με το ΣΥΣ2 και τον ε, οδικό χάρτη που έχουμε για το ΣΥΣ2 δεν θα επηρεάσει τον οργανισμό. Για το θέμα της διαλειτουργικότητας, της ε, διασύνδεσης, φυσικά και κατανοούμε τις ανησυχίες. Δεν είναι μόνο του Κοινοβουλίου και σαφώς δεν θα πρέπει να ποτέ να γίνεται οποιαδήποτε ε, λειτουργική διασύνδεση μεταξύ βάσεων δεδομένων χωρίς απόφαση του ε, Διοικητικού Συμβουλίου και φυσικά αυτή είναι και η λογική μέσα στην οποία φτιάξαμε την πρόταση αυτή. Οποιαδήποτε μελλοντικά συστήματα που χρειάζεται με κάποιο τρόπο να συνδεθούν για λειτουργικού σκοπούς με υφιστάμενα συστήματα θα γίνει αυτό μετά από τη δημιουργία νέας νομικής βάσης για το εν λόγω σύστημα. Άρα λοιπόν έτσι θα υπάρχει δυνατότητα να γίνουν παρατηρήσεις και να κρίνουμε την εγκυρότητα μιας τέτοιας σύνδεσης και διαλειτουργικότητας. Ανάλυση κόστους ωφέλειας και οδικός χάρτης. Αυτό είναι κάτι επίσης που αναφέρθηκε. Για το κόστος ωφέλειας να θυμίσω το γεγονός ότι η αξιολόγηση αντικτύπου έλεγξε εις το θέμα κόστους ωφέλειας για τον οργανισμό καθώς και την καταλληλότητα ενός από τα σενάρια τα οποία εξέτασε η ε, μελέτη αντικτύπου και η σύσταση που υπευλήθη και την οποία ακολουθήσαμε ήταν η πιο οικονομική. Όσον αφορά τον οδικό χάρτη, νομίζω ότι αναφερθήκατε στα οδικού χάρτη του συστήματος. Αυτά δεν θα πρέπει να έχουν επιπτώσεις στην υπηρεσία. ούτε να επηρεάσουν την λειτουργία του οργανισμού. Και όσον αφορά το ΣΥΣ2, ήδη το αντπάντησα, νομίζω. Ευχαριστώ πολύ. Okay, thank you. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κατόπιν αυτή τη συζήτηση για τις τροπολογίες με τον εισηγητή και τους χειόδους εισηγητές, να σας θυμίσω ότι έχουμε μία ψήφο προσανατολισμού στην επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ στις 11 Οκτωβρίου. Αυτά είναι το 10.30 και σχεδόν έχουμε τελειώσει γιατί το σημείο 18 έχει αναβληθεί. Αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντονιστές που συμφώνησαν να αναβάλουν επίσης την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών, των ιδίων για την επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ ώστε να μπορούν να είναι παρόντες όλοι οι συντονιστές. Αν δεν υπάρχει τίποτα στα διάφορα, τελευταία λέξη να σας θυμίσω τις ημερομηνίε για την επόμενη συνεδρίαση της ΛΥΜΠΕ 28 Σεπτεμβρίου. Θα εδώ στις Βρυξέλλες. 3 με 6 με 4,5 και 29 Σεπτεμβρίου. 9 με 12.30 και 11 Οκτωβρίου 3 με 6.30. Σας ευχαριστώ όλους. Where is the meeting this afternoon?